Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με το πρώτο σημείο στην εμμυρική διάταξη, την έγκριση αυτής και να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η ψηφοφορία για τη σχέδια έκθεσης του κυρίου Χέλνερ για την έγκριση τύπου, το σημείο 11 που προβλεπόταν για αύριο, αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της ΕΝΒΗ στις 28. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η μερίσια διάταξη εγκρίνεται ως έχει. Και στο σημείο 3 στις ανακοινώσεις για την ομάδα εργασίας LIFE, η οποία θα λάβει χώρα αύριο στις 8 Νοεμβρίου, από τη 1 ως τις 3, στο, ε, στην αίθουσα 3G2 ASP, με τους υπευθύνους του προγράμματος Live της Γενικής Διεύθυνσης ΕΝΒΗ και ΙΑΣΜΕ. Η συνεδρία είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Σημείο 2. Η ενημέρωση από την ε, συνεδρίαση στη Γερμανία, έκθεση από την από την ε, Regional Fairband Ruhr Essen στη Γερμανία που έλαβε χώρα στις 19 και 21 Σεπτεμβρίου 2016. Έπειτα για την κοινή συνεδρίαση Agri Envy Itre, η οποία θα οργανωθεί στις 21 Νοεμβρίου τη Δευτέρα στο Στρασβούργο για την ε, στρατηγική της δασοκομείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Επίτροπο Χόγκαν. Σήμερα έχουμε διερμενία σε 21 γλώσσες και ως συνήθως Έχετε όλα τα κείμενα στα ηλεκτρονικά σας αρχεία και η συνεδρίαση θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο. Στο σημείο 4. Να θυμίσω ότι έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης 23 και 24 Μαΐου, 21 Ιουνίου, 11 και 12 Ιουλίου και 8 Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις με το τέλος της συνεδρίασης, ε, εγκρίνονται. Περνάμε στο σημείο 5 στην τα ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Χέρτ Ντάνσερτ, τον ε, διευθυντή της ε, ECHA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Ουσιών. Ξέρετε ότι έχουμε διευθυνό διάλογο με τον οργανισμό στα πλαίσια της ετήσιας ανταλλαγής απόψεων και έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού και κυρίω του στρατηγικού του στόχου μέχρι το 2018. Ξεκινώ δίνοντα το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Ντάνσετ και μετά θα έχουμε συζήτηση με τα μέλη τη Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπροεδρία, αξιότιμα μέλη τη επιτροπή, είναι ικανοποίησή μου να είναι εδώ μαζί σα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητα του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Θα προσπαθήσω εισαγωγικά να σα αναφέρω ποια είναι η συνεισφορά του οργανισμού μου σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να δούμε πώ συνεισφέρουμε για να αντιμετωπίσουμε κάποιε από τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και θα αναφέρω και κάποιε προκλήσει ε, εγώ ανυπομονώ να ακούσω τη δική σα ανάδραση και να απαντήσω σε ενδεχόμενε ερωτήσει. Πρόκειται λοιπόν για καιρού προκλήσεων και υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πολιτών, αργεί να ανακάμψει η οικονομία ε, και υπάρχουν ανησυχίε για το κλίμα και για τη ρήπανση. Και εσεί ε, έχετε ένα ζωτικό ρόλο για να απαντήσετε σε αυτές τις προκλήσεις. Κάθε ευρωπαϊκό θεσμό, ε, κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να συνεισφέρει για την εξέβρεση λύσεων. Διαφορετικά είμαστε απλώ τμήμα του προβλήματο Θέλω να εξηγήσω πώ ο δικό μου οργανισμό βοηθά. Αλλά Καταρχήν, ας αναγνωρίσουμε τι πηγαίνει καλό στην Ευρώπη. Καταρχήν, ε, είμαστε επικεφαλείς ε, σε ό,τι αφορά το να έχουμε πιο ασφαλείς χημικές ουσίες ε, και είμαστε περήφανοι. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε ότι η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακίας και θα πρέπει να είμαστε κολακευμένοι που τόσο σε πολλές χώρες παγκοσμίω εμπνέονται από αυτά που κάνουμε στην Ευρώπη για τις χημικές ουσίες. Θα μιλήσω καταρχήν για τη θετική μας συνεισφορά για τους πολίτες της Ευρώπης. Κάνουμε πιο ασφαλή την Ευρώπη. Φυσικά η βελτίωση αυτή δεν γίνεται μία νυχτή. Ενώ το ίδιο το είναι ήταν μια επανάσταση, ο αντίκτυπος του είναι περισσότερο μια εξέλιξη. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο ενθουσιώδες, συναρπαστικό, αλλά το γεγονός είναι ότι πίσω από τα παρασκήνια με αποτελεσματικό τρόπο. Η νομοθεσία που θέσατε σε εφαρμογή πριν 10 χρόνια έχει σημαντικό θετικό αποτέλεσμα στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον για όλους. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς η νομοθεσία του ΡΙΤΣ μας κάνει να είμαστε πιο υγιείς, βοηθά το περιβάλλον και ταυτόχρονα εξοικονομούμε χρήματα. Αφορά το μόλιβδο. Μέχρι πρόσφατα μπορούσε να βρει κανείς μόλιβδο σε προϊόντα όπως ε, σε τυπωμένα τισέρτ, ε, στα φερμουάρ και σε ανακυκλωμένα πλαστικά. Ξέρουμε τώρα ότι η έκθεση στο μόλιβδο μπορεί να βλάψει σοβαρά τον εγκέφαλο και μόνιμα, κυρίως σε παιδιά κάτω των τριών ετών. Τώρα, χάρη στο Ρίτς, η χρήση του μολύβδου περιορίζεται σε τέτοια προϊόντα, δηλαδή 13 εκατομμύρια νεαρά παιδιά δεν εκτίθεται πλέον σε μολύβδο και η ικανότητά τους να μάθουν προστατεύεται και έχουμε έτσι και εξοικονόμηση στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, εκατοντάδες χημικές επικίνδυνες ουσίες τώρα είναι υπό έλεγχο και φυσικά τίθενται υπό όλο και πιο αυστηρό έλεγχο. Οι εταιρείε χρησιμοποιούν την ε, γνώση τους για τις ουσίες, για την παραγωγή πιο ασφαλές των προϊόντων και τη θέση σε εμπορία. Όλο και περισσότερες εμπορίες και κλάδοι της βιομηχανίας αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να εξαλείψουν τις επικίνδυνες ουσίες με δική τους πρωτοβουλία και αυτά είναι πολύ καλά νέα για τους λόγους της Ευρώπης. Η δεύτερη συνεισφορά μας για τους πολίτες είναι η γνώση. Ο Κόφι Ανάν αν είχε και όταν είπε ότι η γνώση είναι δύναμη και η πληροφόρηση απελευθερώνει, τότε το ΡΙΤΣ δίνει επίση δύναμη και απελευθέρωση στου πολίτε μα. Πέρσι σα μίλησα για το βελτιωμένο τρόπο για να ψάξει κανείς ε, ενημέρωση, πληροφορίες για τα χημικά στην ιστοσελίδα μας. Και τώρα χαίρομαι να σας πω ότι από τον Ιανουάριο έχει χρησιμοποιηθεί από δύο εκατομμυρία ανθρώπους. Το χρησιμοποιούν για να μάθουν και τον αντίκτυπο συγκεκριμένων χημικών ουσιών στους ίδιους, στις οικογένειές τους, ε, στους εργαζομένους τους, στους πελάτες τους και στο περιβάλλον. Και αυτή η γνώση έχει αντίκτυπο στις επιλογές που κάνουν. Είναι η πιο πλήρης βάση δεδομένων για τις χημικές χημικές ουσίε παγκοσμίω με δεδομένα ευνόητα για 120.000 ουσίε που διατίθεται ελεύθερα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εργαζόμαστε τώρα και σε μια εκδοχή που θα μπορεί να την κατεβάσει κανεί. Αυτό το σημαίνει ότι οι ακαδημαϊκοί δημοσιογράφοι θα μπορούν να αναλύσουν και να συγκρίνουν τα δεδομένα με δημιουργικού τρόπου και έτσι αυτό θα προωθήσει τη γνώση και την προστασία. Επιπρόσθετα, τώρα που έχουμε δεδομένα που είναι πιο χρήσιμα στους πολίτες. Εργαζόμαστε για μια νέα ιστοσελίδα, ειδικά για αυτούς. Θα περιλαμβάνει και πληροφορίες για τα ανανοηλικά, όπως ξέρετε, η Κομισιόν μαζί ζήτησε να φιλοξενήσουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ανανοηλικά και με τους υφιστάμενους πόρους θα βάλουμε δυνατά μας για να δώσουμε στους καταναλωτές αξιόπιστες πληροφορίες για τα ανανοηλικά στα οποία μπορεί να εκτίθενται. Οι πολίτες ε, απευθύνονται ε, όλο και περισσότερο στον οργανισμό μας απευθείας με τις ε, ανησυχίες τους. Είναι κάτι που εκτιμώ και φαίνεται ότι εκτιμούν τι κάνουμε και τις, εκτιμές που τους, και τις συμβουλές που τους δίνουμε. Τα πιο καυτά θέματα δεν θα σας εκπλήξουν. Το πρώτο είναι το γλυφοσάτ. Ε, οι πολίτες μας όθησαν να κάνουμε μία πλήρη ανάλυση της ταξινόμησης της ουσίας, καθώς κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι καρκινογόνος. Ήμασταν ανοιχτοί με τους πολίτες, ε, τους εξηγήσαμε την αρμονισμένη διαδικασία ταξινόμησης, δημοσιεύσαμε τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων, είχαμε μια δημόσια διαβούλευση και οργανώσαμε παρουσιάσεις από τους κύριους πρωταγωνιστές ε, στη συνάντηση της Επιτροπής στο περίμενα μήνα, όπου θα εξεταστεί για πρώτη φορά η ουσία. Ελπίζω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Κινδύνου θα μπορέσει να γνωμοδοτήσει για το κλειφωσάτ πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι η δοκιμή χημικών στα ζώα. Οι πολίτες ε, θέλουν να σταματήσει αυτό ή τουλάχιστον να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Όπως ξέρετε δεν είναι δυνατόν να το σταματήσουμε εντελώς μέχρι να έχουμε εναλλακτικέ, ε, όπως πρέπει χάρη να δούμε αν είναι καρκινογόνα ή τοξικά ε, αυτά τα προϊόντα. Όμως θέλουμε να διατηρήσουμε ως δυνατόν το ελάχιστο της δοκιμές στα ζώα, δίνοντας συμβουλές στις εταιρείε και απαιτώντα από τις εταιρείε να εξετάσουν αυτές τις εναλλακτικές πριν να ζητήσουν δοκιμές στα ζώα. Ανυπομονώ να λάβει χώρα το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες η διάσκεψη της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που τόνισα στην αρχή αυτής της ακρόσης ε, ήταν η αργή οικονομική ανάκαμψη. Οι βιομηχανίε των χημικών και των μετάλλων είναι θεμελιώδεις για την οικονομία μας ε, σε ό,τι αφορά το εισόδημα που δημιουργούν, αλλά κυρίως ε, επειδή αποτελούν τη βάση όλης της ευρωπαϊκής μεταπητικής βιομηχανίας. Ένας τομέας χημικών ουσιών που θα λειτουργεί καλά και θα παράγει υλικά των οποίων οι κίνδυνοι είναι κατανοητοί και ελέγχονται οι κίνδυνοι είναι ζωτικοί για όλο τον μεταπητικό τομέα. Ε, η χρήση τους έχει βασική οικονομική έννοια, αλλά επειδή θα έχουμε και αποτελέσματα σε πιο πράσινα προϊόντα. Επιπλέον, ε, ουσιαστικά ενθαρρύνουμε τις καινοτόμες εταιρείες να βρουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές Μία πρόσφατη μελέτη ε, από Αμερικανούς ακαδημαϊκούς ε, βρήκε ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ουσιαστικά οδηγεί σε πιο αποτελεσματική αντικατάσταση των χημικών ουσιών στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική πάνω από 1500 νέα και πιο πράσινα χημικά έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησε το ΡΙΚΣ. Αναγνωρίζει η βιομηχανία ότι πρέπει να καινοτομήσουμε και να φέρουμε νέε ιδέε στην αγορά πιο γρήγορα. Γι' αυτό βοηθά το ΡΙΤΣ, μειώνοντα τι νομικέ απαιτήσει σε χημικά που τίθενται ε, στο εμπόριο και τα χημικά που χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη. Όμω πρέπει να έχουμε και ένα feedback ε, από τον κλάδο σε σχέση με το κόστο και το φορτό εργασία τη συμμόρφωση με το ΡΙΤΣ. Αυτό φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο για εταιρείε που ζητούν αδειοδότηση να χρησιμοποιήσουν μία εσύ υψηλή ανησυχία και για μικρέ εταιρείε που εγγράφουν ουσίε με χαμηλού όγκου παραγωγή. Εργαζόμαστε σκληρά με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ε, προκειμένου η συμμόρφωση να είναι όσο δυνατόν ε, πιο εύκολη ε, και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλίσουν οικονομική και άλλη υποστήριξη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τι μικρότερε εταιρείε. Η μόρφωση είναι προ το όφελο όλων. Και έρχομαι τώρα σε ένα σημαντικό σημείο που αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, όπου μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε έχουν επενδύσει πολύ χρόνο και χρήμα στο ε, να παράσχουν τις πληροφορίες που απαιτείται από το ΡΙΤΣ για τις ουσίες που παράγουν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ουσιαστικά να προ υπάρξουν αποτελέσματα των επενδύσεων αυτών και για να έχουμε δηλαδή πιο ασφαλή χημικά, αλλά και για να πληρούνται οι νομικές υποχρεώσεις. Ε, το... Δεδομένα που δημιουργούνται για το ΡΙΤΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την προστασία των εργαζομένων, για την ποιότητα του αέρα και του νερού κτλ. Έτσι θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα κάνουμε τη συμμόρφωση λιγότερο δαπανηρή και πιο αποτελεσματική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη, το REIT σίγουρα έχει ένα κόστος, όμως δίνει και όθηση μεγάλη στην καινοτομία και το πραγματικό τρίκ θα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα κεφαλοποιήσουμε τις επενδύσεις που γίνονται στην ασφάλεια από τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Το τρίτο θέμα που ανέφερα στην αρχή ήταν η ανησυχία για το κλίμα και η ανάγκη να έχουμε ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Τα δεδομένα μας βοηθούν να οικοδομήσουμε την εικόνα για τον αντίκτυπο που έχουν οι χημικές ουσίες στο περιβάλλον. Φυσικά τα χημικά είναι ουσιαστικό τμήμα της κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορεί να υπάρχει κυκλική οικονομία αν δεν υπάρχει καλύτερος έλεγχος και ευαισθητοποίηση για τα πιο επικίνδυνα χημικά. Αν υπομονούμε να υποστηρίξουμε στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτό το τομέα, μπορεί να γίνει ένα ακόμα παράδειγμα ηγετική θέση στην Ευρώπη, στον κόσμο και η πρόκληση θα είναι η Κομισιόν να υλοποιήσει τα φιλόδοξα σχέδια και με τη βοήθεια φυσικά και οργανισμών ε, που θα αναφέρω στις δικές σας επιτροπές Τώρα, ε, θέλω να αναφέρω τρεις προκλήσεις. είναι στο τελευταίο του θητείας μου και έχω εμπνευστεί από τον πρόεδρο Ομπάμα και πραγματικά θέλω να πω ότι τρέχω σε μια σκητελοδρομία και θέλω να περάσω τη σκητάλη μου ε, στο διάδοχό μου και να του δώσω ένα προβάδισμα. Τρία πράγματα έχω κατά νου. Καταρχήν η προθεσμία καταγραφής για το ρίτσο 2018. Να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντικό είναι. Μόνο όταν αυτή η προθεσμία θα γίνει σεβαστή επιτυχώ. θα έχουμε αυτό που απαιτεί το REACH, πλήρη γνώση για όλες τι χημικές ουσίες στην ευρωπαϊκή αγορά σήμερα. Οι εταιρείε θα εγγράψουν πολλά περισσότερα χημικά για αυτή την τελική ημερομηνία από ό,τι ποτέ πριν και τις ουσίες που γίνονται μόνο, παράγονται μόνο κατά ένα τόνο ετησίας. Όμω, ανησυχώ για το ότι πολλέ εταιρείε δεν γνωρίζουν ακόμα τι ευθύνε του και Άλλε έχουν αποφασίσει να μην προβούν στην καταγραφή, αλλά δεν το λένε στους πελάτες τους. Αυτό θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα στους πελάτες που βασίζονται στις εταιρείε αυτές για τα χημικά που χρειάζονται. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα. Οι παρασκευάστρε εταιρείε θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα χημικά που χρειάζονται και παρέχονται σε χαμηλού όγκου εγγράφονται από του προμηθευτέ του και αν χρειάζονται βοήθεια θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή μαζί μα. Το δεύτερο που με ανησυχεί είναι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα με την ποιότητα των δεδομένων για πολλέ από τι χημικέ ουσίε που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Περίπου τα δύο τρίτα όλων των φακέλων που έχουμε εξετάσει μέχρι σήμερα έχουν ανεπαρκή δεδομένα και αυτό σχετίζεται κυρίω με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τη χημική ουσία. Αυτά τα φτωχά δεδομένα μα αφήνουν ουσιαστικά στο σκοτάδι σε σχέση με του πραγματικού κινδύνου ε, που διατρέχουμε αν χρησιμοποιούμε επικίνδυνε ουσίε. Εμεί και τα κράτη-μέλη επικεντρωνόμαστε σε φακελού όπου έχουμε σοβαρή ανησυχία για κάποια χημική ουσία και όπου οι επιπτώσει θα μπορούσαν να είναι σοβαρέ. Όμω πρέπει αυτό το πρόβλημα να επιληθεί ε, αν χρειαστεί με δοκιμέ στα ζώα και δεν μπορούμε να, να βασιστούμε ε, μόνο στην επίσημη διαδικασία λήψη αποφάσεων, καθώ είναι αργή, πρέπει να δεσμευτεί ο κλάδος ότι θα παράσχει δεδομένα ποιοτικά για τις ουσίε, στα πρότυπα του Και το τρίτο είναι η αναθεώρησή μα για τη διαδικασία έγκριση και ιδίω ο ρόλο των επιτροπών μα, το να λάβουμε υπόψη του κοινωνικονομικού παράγοντε στη λήψη αποφάσεων. Εσείς ε, με το ψήφισμά σας της 25ης Νοεμβρίου 2015 προδοτήσατε αυτή την ε, νομοδότηση από τότε εμείς με τη βοήθεια του Διοικητικού μας Συμβουλίου έχουμε προβληματιστεί επί των κριτικής που κάνετε και έχουμε λάβει για κάποια πρακτικά μέτρα. Είχαμε μία καρποφόρο συζήτηση με την Κομισιόν, μέλη του Κοινοβουλίου και τα διαφορεμένα μέρη τον Ιούνιο για τον υποστηρικτικό ρόλο που παίζει η, η κοινωνική οικονομική ανάλυση στην διαχείριση κινδύνου. Από πρακτική σκοπιά παράγουμε ένα πρακτικό οδηγό για τις εταιρείε που θα έπρεπε να οδηγήσει σε καλύτερες ε, ε, αιτήσει για την ποιότητα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία. Και ουσιαστικά να δούμε τι γίνεται με το σε ποιο ασφαλείς εναλλακτικέ που υπάρχουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα. Και μαζί με την Κομισιόν εργαζόμαστε για μια διαδικασία για τα αντιαλλακτικά και για τις ουσίε χαμηλού όγκου. Επίσης, ε, θέλουμε να παράξουμε γνωμοδοτήσεις πιο κατανοητές και συνεκτικέ. Συζητούμε την πρόοδο με το Διοικητικό μα Συμβούλιο το Δεκέμβριο και θα επανέλθουμε σε εσά γραπτός. Σας ευχαριστώ και πάλι που με προσκαλέσατε να απευθυνθώ σε σας εδώ και σας ευχαριστώ για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον στο έργο μας και φυσικά και για τη βοήθειά σας στο να διατηρήσουμε και τις, τους πόρους εμπειρογνωμοσύνης μας τον επόμενο χρόνο. Θα ήθελα να εκφράσω και το θαυμασμό μου προς την κυρία Τζούλη Γκίλινγκ, η οποία στη δέσμευση και η κατανόηση ήταν παραδειγματική. Χαίρομαι που ακούω ότι θα καλωσορίσουμε στο Ελσίνκι του χρόνου μία αποστολή από την Επιτροπή και ελπίζω να δω κάποιους από εσά και το προσωπικό σας σε μια σύντομη ενημέρωση που θα δώσει αύριο η Τζούλη στο Κοινοβούλιο αύριο το πρωί. Ελπίζω ότι θα θεωρήσετε ότι είναι χρήσιμο να έχετε μια καλύτερη εις βάθος ματιά της ε, σημερινής μας εργασίας. Σας ευχαριστώ και πάλι και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το υπεύθυνο για τις επαφές μας με, την, τον οργανισμό. Τζούλη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας ε, λόγια. Δεν θα κάνω ανασκόπηση και δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες όλες σας τις παρουσίασης, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη και νομίζω κάλυψε τα βασικά σημεία. Ήθελα απλώς να θίξω ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μου επισημάνθηκε από αρκετούς ενδιαφερομένους φορείς και των εταιριών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό έχει να κάνει με τη διάθεση πληροφοριών. Και το θίξατε κάπως στην ομιλία σας και εσείς. Το θέμα είναι ότι αρκετοί οργανισμοί μεταξύ των οποίων και εσείς και η ΕΜΑ και η ΕΦΣΑ ε, συλλέγεται παρόμοιο είδους πληροφορίες. Και ιδίω όπω συνεχίζουμε εμεί τη σχετική μελέτη με του ενδοκρινικού διαταράκτε, οι πληροφορίε συσσωρεύονται. Το πρόβλημα είναι λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διαφοροποιήσουμε την συλλογή πληροφοριών. Διότι το να συλλέγουν με παρόμοιο, κοντινό τρόπο οι διάφοροι οργανισμοί παρόμοιε πληροφορίε ανάλογα με την εσωτερική αρμοδιότητα και πολιτική του κάθε οργανισμού, τις ανάγκες των εταιριών, τέλο πάντων οτιδήποτε εκπροσωπούν, ε, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εάν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί συμφωνούσαν να έχουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση στα δεδομένα, ιδίω στα δεδομένα ασφαλεία, όπου υπάρχουν ε, φοβερέ ε, ανησυχίε από το κοινό και φοβερή προσοχή για τι δοκιμέ σε ζώα, λόγω χάρη. Ε, με το πρόγραμμα REACH έχουν αυξηθεί οι δοκιμέ στα ζώα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που έχει επικρατήσει. Άρα με όσα συμβαίνουν και επειδή υπάρχουν και εθνικέ ρυθμιστικές αρχέ που έχουν τις δικές τους, ε, τη δική του συλλογή πληροφοριών, το ίδιο και οι εταιρείε και επιχειρήσει επιχειρήσεις, σε αυτή την ε, φάση λοιπόν, θα ήταν καλό νομίζω να ζητούσαμε από τους οργανισμούς μας να έχουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση Μάλιστα, θα πρέπει να γίνει αυτό επισήμω και η Επιτροπή μα να έχει σε αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο καλύτερο τρόπο θα ήταν ίσω να οργανωθεί μια ακρόαση όπου όλοι οι οργανισμοί και οι τρει να συμμετέχουν και να υπάρξει μια συζήτηση έστω και ανεπίσημη για να σχεδιάσουμε κάτι για το μέλλον. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν συμφωνείτε να γίνει κάτι τέτοιο και αν θα μπορούσε να εμπλακεί πλήρω ο οργανισμό σα σε μια τέτοια διαδικασία εφόσον εγκριθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο αντιπρόεδρος κύριος Ποτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω κύριε Ντάσετ γιατί θαυμάζω ε, το έργο σας Θυμάστε πέρσι το Κοινοβούλιο ανέκρινε ένα ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία για τα ανακυκλωμένα ε, πλαστικά. Και παρά ε, τα μεγάλα προβλήματα και το σαφή κίνδυνο για τις εργαζόμενες οι γυναίκες κυρίως, ε, το θέμα αυτό συζητήθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για τα Χημικά και με διάφορες ε, άλλες οργανώσεις και φορείς. Σας ευχαριστώ για τη θετική σας ε, στάση απέναντι σε αυτό το θέμα, αλλά ε, να σας κάνω και μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Τώρα που βρισκόμαστε με τις επιτροπές της, του ΕΚΑ, θα αλλάξουν την πρακτική τους και θα τους ενθαρρύνεται να απορρίπτουν τις αιτήσει ε, γραφής ε, όταν αυτές δεν είναι ε, σωστά διατυπωμένες ή αναποτελεσματικές. Ευχαριστώ κύριε Ντάλ. Ευχαριστώ κύριε Ντάσετ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να αφαιρθώ στον κατάλογο 117 ουσιών για το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2017-2019 που έχετε γράψει σε ένα κατάλογο αυτό. Υπάρχουν πολλές ουσίες που πρέπει ε, να ε, ελέγχονται κάθε χρόνο και του χρόνου ε, πρόκειται να εξετάσετε μόνο 24 ουσίες που είναι αριθμός πολύ χαμηλότερος από εκείνον των προηγούμενων ετών. Αλλά για να αρχίσει η εξελόγηση χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Θέλω να σας κάνω ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες. Πώς μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε ότι δεν θα ε, ανταμείβεται τις εταιρείε που θα έχουν ε, μη ολοκληρωμένο φάκελο όταν πρέπει να ελεγχθεί η ουσία. Και μάλιστα μέχρι και τέσσερα χρόνια πριν αρχίσει η αξιολόγηση. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα στόχο το 2020 να υπάρχει ένας κατάλογος με ε, στοιχεία ουσιαστικά, αλλά χρειάζεται να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Από την άλλη όμως, κινδυνεύει αυτό να οδηγήσει σε ένα ε, μποτιλιάρισμα, ας πούμε σε μια συσσόρευση ε, επικινδύνων ουσιών. Ας εσείς αυτό το θεωρείτε πρόβλημα και πώς πιστεύετε ότι θα φτάσετε στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμέσμακερ Μάκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ε... Εδώ κάθομαι κιόλας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Ντάσετ. Στην εισαγωγή σας μιλήσατε ακριβώς για την κυκλική οικονομία. Και ρωτώ, γιατί εγώ είμαι σκιώδης ηγητής, ξέρετε, ε, ε, από την ομάδα ICR e των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Και έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχει το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία που μεταξύ άλλων θέλει να τονώσει την ανάπτυξη μιας αγοράς ή πολλών αγορών για δευτερογενείς πρώτες ύλες. Βλέπε χημικά, γιατί εκεί εντάσσονται τα χημικά γιατί υπάρχουν ορισμένες ουσίες που μπορεί να είναι, να μην είναι επικίνδυνες και να ε, ανακυκλώνονται. Στο πρόγραμμα δράσης προβλέπεται για το 2017 και παραθέτω μια ανάλυση και πολιτική στα πλαίσια της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα και ε, τα απόβλητα, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο η παρουσία ανησυχητικών ουσιών στα προϊόντα μπορεί να μειωθεί και να βελτιωθεί η χνηλασιμότητα. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε στην εισαγωγή σας ότι θέλετε να δείτε τι ρόλο μπορείτε εκεί να διαδραματίσετε. Τι ακριβώς εννοείτε. Τι ρόλο δηλαδή θέλει να παίξει ο οργανισμός σας αυτή τη διαδικασία. Είμαι περίεργος να μάθω τις συζητήσεις που έχουμε. Ε, να μας πείτε και ποια είναι η άποψή σας. Πώς έχει η προεργασία που γίνεται ακριβώς για αυτή όλη την προσπάθεια της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μέλιορ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από πλευρά μου τον κύριο Ντάνσετ για αυτά που μας είπατε και σήμερα αλλά και συνολικά το έργο σας γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος ε, που έχετε να διεκπαιρεώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας προσωπικά φυσικά και τους συνεργάτες σας άνδρες και γυναίκες. Έχω δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη ο Επίτροπος Ανδριοκάητης εξήγηλε ότι θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τις ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Και εκεί ε, ο δικός σας οργανισμός ε, για τα χημικά παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Είστε προετοιμασμένοι να τον αναλάβετε αυτό το ρόλο, σας έχει προβληματίσει ήδη πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων και η προετοιμασία. Και ερώτηση δεύτερη. Αναφερθήκατε σύντομα στο πρόβλημα των πειραμάτων με ζώα. Γνωρίζουμε ότι στην έρευνα γίνεται μεγάλη πρόεδρος, πρόοδος συγγνώμη, με καλλιέργεια ιστών, ε, όπου μπορούμε να δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα και να γίνουν διάφορα πειράματα. Ερώτηση. Ποιο μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να φύγουμε από τα πειραματόζωα και να πάμε σε ιστούς που θα έχουμε καλλιεργήσει ε, στο εργαστήριο για να μην έχουμε καθόλου πειραματόζω. Κανονικά αυτό θα ήταν μια διαδικασία ταχύτερη και φθηνότερη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πειραματόζω, υπάρχουν και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ. Κύριε Ντορνανό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Διευθυντά, για την ε, προσοχή σας. Εγώ ήθελα να σταθώ στα φυτογειονομικά προϊόντα. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού του 1991 για τη βιολογική καλλιέργεια για τις βιολογικές καλλιέργειες ε, του 2000, ε, που τροποποιεί τον κανονισμό του η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα θέσουν ένα νέο πλαίσιο για τη χρήση των φυτογενομικών προϊόντων. Όμω οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Γεωργία έχουν ήδη εδώ και δύο μήνε ε, δείξει ανοχή σε ένα ποσοστό χημικών ουσιών σε φυτοφάρμακα και μη γενετικώ τροποποιημένου σε κάποιε βιολογικέ καλλιέργειε. Ο λόγο είναι για να προωθηθεί καινοτομία, ανταγωνιστικότητα αλλά και η προστασία τη ε, ανθρώπινη υγεία καθώ και το περιβάλλον. Γι' αυτό ήθελα να σας ε, καλέσω και να σας, να, σας ρωτήσω μάλλον και να ζητήσω πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος ξεκινώντας να υποβαθμίζουμε τα πρότυπα. Πρώτα απ' όλα θα πληγεί η, ποιότητα των προϊόντων με την ε, φυτογεωνομική τους ε, σύσταση. Γιατί να επιβληθούν ποινές σε καλλιέργειες που έχει τετραπλασιαστεί η ανάγκη για την Επίσης με ένα δίκτυο εμπιστοσύνη 80% βάσει των μελετών μιας Γαλλικής Ένωση Καταναλωτών, τα βιολογικά προϊόντα θα χάσουν ένα μεγάλο μερίδιο της του τους ε, στα μάτια των καταναλωτών με μια τέτοιου είδους απόφαση. Και εν τέλει οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις θα υποφεληθούν ει βάρο των ε, ε, σε ανθρώπινε διαστάσει εκμεταλλεύσεων. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι Πότε θα λάβετε υπόψη τα στοιχεία αυτά στα πλαίσια του νέου κανονισμού που προτείνεται, διότι εδώ διακυβεύεται η υγεία, αλλά και η επιτακτική ανάγκη να μην ε, υποβαθμιστεί ολόκληρη η γεωργική παραγωγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω αν άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ε, Τώρα μπορούμε να σας δώσουμε χρόνο για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους. Να ξεκινήσω ή μάλλον θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά με την οποία τα έθηκαν οι ερωτήσεις. Ξεκινώ με την ερώτηση για ένα ενιαίο μορφότυπο, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τις πληροφορίες ασφαλείας, τα δεδομένα ασφαλείας, από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων οργανισμών. Να τονίσω ότι μας ενδιαφέρει πολύ να συμμετάσχουμε σε αυτού του είδους ε, την προσπάθεια και ήδη έχει επιτευχθεί σχετική πρόοδος κυρίως στη συνεργασία μας με την ΕΦΣΑ για, τις, ε, για τα φυτογενομικά προϊόντα, τα φυτοφάρμακα. Την αναθεώρηση του πλαισίου για τις ενεργές ουσίες στα συστατικά των φυτοφαρμάκων και τα προϊόντα που τις περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες. Έχει επιτευχθεί λοιπόν πρόοδος για να καταλήξουμε σε μια νέα προσέγγιση για την υποβολή των πληροφοριών από τα κάτι μέλη. Έχουν γίνει και επιστημονικές μελέτες και μελέτες από την πλευρά των εταιριών και επιχειρήσεων για τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα. Και εδώ πιστεύουμε ότι η παρουσίαση βάσει του συστήματος του Euclid είναι ο καλύτερος τρόπος για την εναρμόνιση της συλλογή πληροφοριών. Με την περίληψη των μελετών, την επισκόπηση που είναι ο καλύτερος τρόπος να συγκεντρώνονται τα πορίσματα. Ναι, μας ενδιαφέρει να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία από πλευρά σα. Σε σχέση με το ψήφισμα που εγκρίνατε πέρυσι, για μια αίτηση έγκριση, μια από τι πρώτε, για το DHP στα ανακυκλωμένα υλικά, ναι, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Και όπως είπα, τη σχετική πρόοδο θα τη συζητήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο να απαντήσουμε γραπτός στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Η συνάντηση του Συμβουλίου που θα συζητηθεί το θέμα αυτό είναι το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το όριο των ε, εισερχομένων πληροφοριών χωρίς να επηρεαστεί το κόστος. Θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης να συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και το βαθμό πληρότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε. Επίσης, βάσει της νομοθεσίας, όταν δεν είναι αρκετά ποιοτικέ οι πληροφορίες ώστε να κλείσει το θέμα και να δοθεί μια απάντηση στον Ετούντα για να ε, βελτιώσει τις πληροφορίες του, τότε αυτό πολλές φορές παραμεινεύεται. Λες και βοηθούμε τους Ετούντες και κάνουμε τη δουλειά εκ μέρους τους. Τους υποκαθιστούμε. Δεν ευσταθεί αυτό. Δεν κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν εκείνοι. Απλώς οι επιτροπικοί και εισαγητές της θα πρέπει να διατυπώνουν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις ώστε να δίνουμε και μια τελευταία ευκαιρία στον Ετούντα. Είναι σαφές στο νου μας ότι εάν ο ετών έχει δώσει τις πληροφορίες, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ε, διαμορφώσουμε μια ε, τεκμηριωμένη άποψη, κάτι, κάποια λύση πρέπει να δοθεί. Για τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός τους, πρέπει να πω, λόγω της ανάγκης του πρώτερου, της δοκιμής πρώτερης ε, συμμόρφωσης που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν μπουν στον κατάλογο. Βάσει του, των αποφάσεων του εφετείου. Η αξιολόγηση των ουσιών έχει καταλήξει να είναι η απέτηση για την υποβολή των βασικών πληροφοριών Δηλαδή συνήθω ζητούνται οι επιπλέον και λείπουν οι βασικέ. Γι' αυτό έχει μειωθεί τόσο πολύ ο αριθμό των ουσιών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και θα παραμείνει χαμηλό αυτό ο αριθμό. Μόλι η έλεγχη συμμόρφωση των ουσιών που έχουν ανακοινωθεί προηγουμένω, το προηγούμενο βαθμολόγιο τη περσινή χρονιά, και μόλι έχουν ληφθεί σχετικέ αποφάσει και έχουμε συγκεντρώσει και τι απαραίτητε πληροφορίε, τότε μπορούν να κάνουν το του αξιολόγηση στα κράτη-μέλη πώς αποφεύγεται η χαμηλή ποιότητα στις εισερχόμενες πληροφορίες. Έχουμε αλλάξει αυτό που κάναμε συνήθως. Δεν επαφιόμαστε πια μόνον στο σύστημα ελέγχου ποιότητα των υπολογιστών για τα διάφορα ντοσχέ, τους φακέλους υποψηφιότητας, αλλά κοιτάζουμε και στο χέρι της αιτήσει. για να είμαστε βέβαιοι ότι στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει έλεγχοι, δεν υπάρχουν αποτελέσματα δοκιμών, είναι τεκμηριωμένη η αιτιολόγηση. Αυτό που θα συζητήσουμε σύμπτωμα με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο Συμβουλίου είναι εάν η δυνατότητες που έχουν διατεθεί στα κράτη-μέλη σε τρία επίπεδα μπορούν να επιτρέψουν σε συνδυασμό να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα με μία ε, μορφή συνεργασίας ε, όλων και με τις εταιρείες και με ε, μια διάθεση θελοντική. Θα τα συζητήσουμε με τα κάτι μέλη τον ερχόμενο μήνα και θα ληφθούν αποφάσει σχετικά στι αρχέ τη επόμενη χρονιά. Με την ε, οικειοθελή προσφορά των κρατών μελών και των εκπροσώπων των ε, εταιριών. Για να μην περιμένουμε τι τελικέ αποφάσει προκειμένου να βελτιώσουν ε, τα ντοσιά του φακέλου του. Αυτά επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή. Ω προ τι ερωτήσει για την κυκλική οικονομία. Ναι, Συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τους εκπροσώπους της Επιτροπής το πρώτο εξάμεινο της φετινής χρονιάς. Για το πώς μπορούμε να τους διευκολύνουμε ώστε τα σχετικά πολιτικά έγγραφα να είναι πιο συγκεκριμένα. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο, την ανάλυση των πολιτικών επιλογών. Αυτό όντως θα ήταν ε, σημαντικό ώστε οι ουσίες που απασχολούν πολύ δεν ανακυκλώνονται και ξαναμπαίνουν τελικά στο σύστημα. αν υπομονούμε να κάνει συγκεκριμένε προτάσεις η Επιτροπή. Για να τοποθετηθούμε κι εμείς όπως είχαμε συμφωνήσει. Έτσι είχαμε πει να προχωρήσουμε. Για την ώρα όμω δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση, κανένα σχέδιο πρόταση, οπότε δυστυχώ. Θα υπάρχει πρόκληση. Τα σχόλια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα κριτήρια. έχουν προβλεφθεί και για τα ζυζανιοκτώνα και για τα παρασυτοκτώνα προτάσεις και θα συνεργαστούμε με την ΕΦΣΑ για να αναπτύξουμε τις κατάλληλες κατευθυντηρίες γραμμές. και να παρακολουθήσουμε στενά και με ιδιαίτερη προσοχή την συζήτηση για τις πολιτικές επιλογές που γίνεται. Και πρωτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κάνει τις τελικές της προτάσεις. Μας πει ποια είναι τα τελικά κριτήρια που επιθυμεί. Θα φροντίσουμε επιστημονικά να στηρίξουμε αυτή τη δουλειά. Ε, όποτε συναντιόνται τα κράτη-μέλη θα το συζητάμε και σε δεύτερη φάση σκοπεύουμε να Έχουμε μια κοινή προσέγγιση για περαιτέρω κατευθυντήρες γραμμέ και για τα ζυζανιοκτώνα και για τα παρασιτοκτώνα. Για τα διοκτώνα και τα παρασιτοκτώνα. Ε, το σημαντικό είναι να υπάρξουν κριτήρια και μια ουσία που έχει μπει στην κατηγορία του ενδοκρινικού διαταράκτη, είτε στα βιοκτώνα είτε στα παρασιτοκτώνα, να είναι ε, γνωστή ως τέτοια, γιατί πολλά χημικά έχουν διαφορετικές χρήσεις ταυτόχρονα. Και τέλος για την ε, πολιτική μας για τα φυτογειονομικά. Δεν μπορώ να σα δώσω κάποια ικανοποιητική απάντηση, διότι ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη μα γι' αυτό. Έχει αυτό να κάνει περισσότερο με τα παρασιτοκτόνα και είναι ευθύνη της ΕΦΣΑ να απαντήσει σε αυτού του είδους τις πολιτικές ερωτήσεις. Βεβαίως, Εάν μας ζητηθεί αυτό θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την ΕΦΣΑ, αλλά νομίζω αυτό αρκεί ως απάντηση. Επίσης, για τις ε, δοκιμές για τα πειράματα σε ζώα και την ερώτηση που θέσατε, ξέχασα να απαντήσω. Εδώ βλέπουμε να οδεύουμε προς το τέλος των δοκιμών σε ζώα. Έχουμε καταφέρει σημαντική πρόοδο ώστε τα in vitro, ε, τα in vitro πειράματα και άλλου είδους δοκιμές για πολλές χημικές ουσίες να γίνουν αποδεκτά. Μακροπρόθεσμα βεβαίως. Οι συνέπειες των χημικών ουσιών και το κατά πόσον θα είναι επικίνδυνες ή όχι είναι κάτι που δεν μπορούμε να, το δούμε, να το δούμε από σήμερα με τις τωρινές Και δεν ξέρουμε αν ιδιότητε που σήμερα ε, βλέπουμε στα πειράματα μπορούν να επιβεβαιωθούν και για το μέλλον. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε το κατά πόσο είναι αποδεκτά αυτά που ήδη γίνονται στις δοκιμές των ζώων και στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα δούμε κατά πόσο η επιστημονική μας γνώση μας έχει εξυπηρετήσει στο να στραφούμε σε άλλες εναλλακτικέ. Του χρόνου δηλαδή θα μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τα πορίσματά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Μπάς, πολύ σύντομα. Μια συμπληρωματική ερώτηση. Μπορεί να έχασα κάτι γιατί καθυστέρησα και ζητώ συγγνώμη. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι τα δύο τέταρτα των αιτήσεων ε, δεν είναι πλήρης. Έτσι, μιλούμε για την ποιότητα των ε, στοιχείων που σας στέλνουν. Τα δύο τρίτα λέτε. Ταυτόχρονα μας λέτε ότι μέχρι τα τέλη του επομένου έτους, και είναι σημαντικό να έχει γίνει μέχρι τότε αυτή η δουλειά, προβλέπεται να γίνει. Αλλά τώρα δέκα χρόνια παραμένει έτσι η κατάσταση, να μην είναι πλήρη τα δύο τρίτα των φακέλων. Και τι μέτρα σκέφτεστε να λάβετε για να πιέσετε έτσι ώστε να σα στέλνουν τα σωστά στοιχεία και επαρκή αυτά που απαιτούνται. Γιατί πολύ σκληρά τα λόγια σα, αλλά δεν ακούω συνέπειε. Και αν παραμείνουν δηλαδή ελλειπή τα στοιχεία, εσεί τι θα κάνετε είναι ότι δεν είναι πλήρη η φάκελοι, αλλά δεν συμμορφούνται. Ένα σχόλιο του μικροφώνου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε την ποιότητα των δηλώσεων, γιατί πολύ συχνά ο κλάδος δεν έχει κάνει αυτές τις μικροπρόθεσμες δοκιμές. Και υπάρχουν δυνατότητες στην νομοθεσία και καθοδήγηση που μας επιτρέπουν να μπορούμε να αποδείξουμε επιστημονικά γιατί δεν χρειάζονται αυτές οι δοκιμές για συγκεκριμένες ουσίες. Και αν αυτή η λογική δεν γίνεται αποδεκτή από τους δικούς μας επιστήμονες, τότε ουσιαστικά λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις αξιολόγησης για να ζητήσουμε δοκιμές ή για καλύτερες εναλλακτικέ για τις δοκιμές. Γιατί ακόμη και όταν παραγγέλνουμε μια δοκιμή, Βασικά, καλούμε τον κλάδο να μας παρουσιάσει ένα καλύτερο αντιπιχείρημα που να ισχύει επιστημονικά, τότε αν ισχύει κάτι τέτοιο μπορούμε να το δεκτούμε. Αυτό ήθελα να το αποσαφηνίσω. Η πολιτική λοιπόν που ακολουθούμε συνίσταται στο εξής. Επικεντρώνουμε την αξιολόγησή μας σε σημαντικές ουσίες, αυτές που ενδυνάμει μπορεί να είναι επικίνδυνες, έτσι ώστε να μην μας απασπάται η προσοχή από σχετικά αθώα χημικά, αλλά να επικεντρωνόμαστε στις ουσίες που ήδη είναι γνωστές ότι έχουν επικίνδυνες ιδιότητες βραχυπρόθεσμα στην υγεία και στο περιβάλλον. Δεύτερον, ανυπομονώ να πετύχουμε μία συμφωνία με κάποιους τομείς εθελοντικά, έτσι ώστε να αποφύγουμε όλη αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατόπιν να έχουμε μία συμφωνία εκούσια προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση σε όλους αυτούς τους φακέλους. Κάτι τέτοιο θα μας εξοικονομούσε πολύ χρόνο. Γιατί αν κάνουμε μία επιτυχή Θεώρηση των δεδομένων, αν κάνουμε δηλαδή καταρχήν ένα τεστ συμμόρφωση, κατόπιν μια επιτυχη θεωρηση τον δεδομενων και κατόπιν μια ανάλυση διαχείριση του κινδύνου και κατόπιν να έχουμε μια πρόταση για περιορισμό ή για ένα μέτρο διαχείρισης του κινδύνου, όλο αυτό διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν να εξελίψουμε όλο αυτό το μακρύ χρονοδιάγραμμα Πώς, αναζητώντας έναν δημιουργικό τρόπο να δούμε πώς με τη μία θα συμφωνήσουμε με τον κλάδο επί όλων των φακέλων και κατόπιν θα συμφωνήσουν μαζί μας σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για να γίνουν σεβαστοί, να συμμορφούνται μάλλον οι Αλλά ε, εσείς ε, μίλησατε τώρα για θελοντικέ προσεγγίσεις, όλα αυτά που ακούγονται κάπω αδύναμα. Αν όχι, τότε θα λάβουμε τι αποφάσει. Ακόμη και αν κάνεις ε, μια εθελοντική δουλειά, αν τελικά ο κλάδο δεν έρθει σε συμφωνία μαζί μα, τότε θα ξεκολουθήσουμε να θα ξεκολουθούμε να εκδίδουμε τις αποφάσεις και μάλιστα θα, κάνουμε... θα εκδώσουμε και μία απόφαση που θα αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και η του χρόνου. Του χρόνου θα κάνουμε μια πιλωτική εφαρμογή για τη δοκιμή. Αυτή είναι η πρόταση. Εδώ τώρα εξετάζουμε διάφορους κλάδους προκειμένου να κάνουμε αυτή τη δοκιμή. Πρόεδρος και η κυρία Σιροπερίκ έχει ζητήσει το λόγο, αλλά τώρα θα κλείσουμε εδώ το κατάλογο των ομιλητών, γιατί έχουμε αργότερα και ένα σημαντικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Κυρία Σιροπερίκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητούσαμε πέρυσι πάρα πολύ στην Ολλανδία. Ξέρετε ότι εδώ είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχουμε την οδηγία για τα νητρικά. Θα πρέπει να χαθούν ε, ε, μισό εκατομμύριο γελάδες του χρόνου από την Ολλανδία. Ε, τι κάνετε για όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς. Εδώ είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εγώ δεν μπορώ να πάω στους αγρότες και να τους πω αυτά που μας λέτε τα γενικά. Πρέπει να τους πω συγκεκριμένα πράγματα. Πώς θα τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά. Κατά την άποψή μου. Εμείς δεν ε, ε, έχουμε αρμοδιότητα για το ΆΙΔΑ. Ε, για το νερό δηλαδή. Υπάρχει οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, για το, τα αζωτούχα, πόσα νητρικά και πόσα νητρόδι μπορούν να περιέχουν τα ύδατα και το πόσιμο νερό. Δεν είναι όμω δική μας αρμοδιότητα αυτό. Τα λέει η ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Δεν αφορά το δικό μας οργανισμό. Θα μπορούσαμε Έχουμε την επιστημονική γνώση και την κατάρτιση. Αν μα ρωτήσουν, συγγνώμη, μπορούμε να απαντήσουν. That, uh, action... Ε, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση όμως σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα. Ε, δεν μπορεί ε, κάποιος να κάνει κάτι, μια δράση ας πούμε, να έχει που να φύγει μόνο τους αγρότες ε, αλλά όχι τη βιομηχανία και το, τα καύσιμα ας πούμε η βιομηχανία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα ε, και ρηπαίνει. Και αυτό συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο οι αγρότες και μπορούν εκεί να ληφθούν επίσης ε, δράσεις. Μπορεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο αρμόδιος αυτός ο οργανισμός, να ε, κάνει προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορεί να είναι στην υπηρεσία σας, ε, ε, η δική μας ε, υπηρεσία, ο οργανισμός μας. Έχουμε πληροφορίες, αρμοδιότητες, όμως δεν έχουμε για κανένα από τα δύο αυτά που ρωτήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ το σημείο αυτό, στη μέση διάταξη και να περάσουμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Ντάνσετ για την παρουσία του εδώ για την πολύ χρήσιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο που είχαμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για την Τρίτη και Τέταρτη Δέσμη. Και τη λειτουργία των συσκευών αναστολής. Η επίμαχη φύση κάποιων στοιχείων των δύο αυτών δεσμών και το θέμα των ε, συσκευών ε, αναστολής που έφερε στο φως το σκάνδαλο του Volkswagen πέρσι μας οδηγεί στο να μελετήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά που προκαλούν τη δημόσια προσοχή και τα μέλη της Επιτροπής εμείς, της Εξεταστικής αυτής Επιτροπής έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν στη σημερινή μας συζήτηση. Ε, να καλωσορίσω, χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω, την κυρία Τζοάννα Σιπόφκα, ελπίζω ότι το πρόφερα σωστά το όνομά σας, που εκπροσωπεί τη Γενική Διεθνή Συγκρόου, και θα έχετε το λόγο για την παρουσίασή σας. Μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μεταξύ των μελών της ε, Επιτροπής μας και των μελών της Επιτροπής εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό Είχαν γίνει και συζητήσει στην αρχή του έτου για το δεύτερο πακέτο για τι δοκιμέ σε συνθήκε πραγματική οδήγηση. Να σα ενημερώσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιε είναι οι προθέσει μα. και με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε έρθει εδώ για να τα συζητήσουμε αυτά μαζί σα για το τρίτο και το τέταρτο πακέτο, Κυρίω το τρίτο γιατί έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος και μπορούμε να σας πούμε σε μεγαλύτερο βάθος τι προθέσεις έχουμε. Ανακεφαλαιώνω. Στόχος ποιος ήταν από την αρχή να κάνουμε ε, δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης ε, σταδιακά και βαθμία. Είχαμε το πρώτο και το δεύτερο πακέτο, το τρίτο που θα σας παρουσιάσω σε λίγο και το τέταρτο το οποίο θα έρθει στις αρχές του επομένου έτους. Όλα αυτά λοιπόν τα πακέτα και οι δέσμες μέτρων ε, θα εγγυώνται ότι θα γίνεται μια σωστή δουλειά με στιβαρή έτσι, μεθοδολογία, με εργαλεία συμμόρφωσης και εφαρμογής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τρίτο πακέτο, έχει να κάνει με τη συμμόρφωση και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας. Είναι τέσσερις κανονισμοί λοιπόν και αυτό ε, θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί του χρόνου, του επόμενους μήνες. Έρχομαι λοιπόν στο λεγόμενο τρίτο πακέτο για τις εκπομπές ε, συνθήκης μαγματικής οδήγησης. Καταρχάς πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Αρχίσαμε στις αρχές του έτους και ήδη το Σεπτέμβριο είχαμε ολοκληρώσει την εσωτερική ανάλυση, είχαμε κάνει τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους κράτη-μέλη, ΜΚΟ, τη βιομηχανία και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοδοξούμε να εγκριθεί πριν το τέλος του έτους. Τι καλύπτουμε λοιπόν σε αυτό το τρίτο πακέτο. Λίγα ε, θέματα που δεν καλύπτονται στο προηγούμενο θα σας ε, αναλύσω στη συνέχεια, αλλά βασικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι μέτρηση των αιωρουμένων σωματιδίων σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Επίσης, έχουμε ε, συμπελάβει την ψυχρή εκκίνηση και ε, ε, συνθήκες πραγματικής οδήγησης για υβριδικά αυτοκίνητα ε, και είναι πάρα πολύ τεχνικά αυτά ίσως που σας λέω, θα τα αναλύσω στη συνέχεια για την αναγέννηση επίσης και για συνθήκες συμμόρφωσης για Ε, για το πιστοποιητικό συμμόρφωση, το Certificate of Conformity ε, και διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ταχύτητες που μετράμε σε μικρά αυτοκίνητα, πολύ μικρά. Και για κατασκευαστές που παράγουν πάρα πολύ λίγα οχήματα. Λοιπόν, ε, γενικά θα σας τα λέω όχι πάρα πολύ ειδικά και τεχνικά, αν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που με βέβαια ότι θα έχετε να σας απαντήσω στη συνέχεια. Πρώτον, ε, για τον αριθμό των ερωμένων σωματιδίων, PN, για ποια αυτοκίνητα μιλάμε, ε, ε, ποιον αφορούν αυτά, τα πετρελαιοκίνητα, δίζελ και πετρέλαιο, Βεβαίω, ο κανονισμό καλύπτει και τα δύο, αλλά ποια είναι η διαφορά, είναι ουσιώδης. Τα διζελοκίνητα ήδη έχουν φίλτρα καταλύτες ενώ ε, τα βενζινοκίνητα δεν έχουν ακόμα φίλτρα ε, για τα ερωμένα σωματίδια, με εξαίρεση ένα ε, τύπο. Ε, ορισμένες εταιρείες, μάλιστα πριν να σε ισχύ αυτό, ε, αρχίζουν και το εφαρμόζουν. Αλλά κυρίως μιλάμε για τα πετρελοκίνητα όταν αναφερόμαστε σε ρούμενα σωματίδια. Στο κοινό κέντρο ερευνών καταλήξαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μετρήσει κανείς σε ορούμενα σωματίδια σε αυτοκίνητα GDI Και σε αντίθεση λοιπόν με τη συζήτηση για τα νόξ, για τα οξύδια του αζότου, μιλάμε για παράγοντα συμμόρφωσης που θα επέτρεπε κάποιο χρόνο ε, ε, για συμμόρφωσης. Ε, τώρα δεν προβλέπουμε ε, κάποια προθεσμία για να συμμορφωθούν οι κατασκευαστές. Διότι υπάρχει η δυνατότητα ε, να το κάνουν αυτό γιατί οι κινητήρες τους ε, έχουν ήδη εξοπλιστεί με ε, φίλτρα καθαρισμού σωματιδίων. Αυτό που μας απασχολεί τώρα λοιπόν είναι να δούμε αν είναι σωστά τα στοιχεία, οι συσκευές μέτρησης δηλαδή για τα ερώμενα σωματίδια έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά ακόμα ε, πρέπει να καλύψουμε ε, τα κενά στην νομοθεσία. Προτείνουμε ένα περιθώριο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ε, καμία παροχή ή υποχώρηση που κάνουμε απέναντι στους κατασκευαστές. Είναι μισό και που προβλέπεται και υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης όσο προχωρούν τα στοιχεία να μειώσουμε αυτό το περιθώριο που του δίνουν. Δεύτερο σημαντικό, η ψυχρή κίνηση, το λεγόμενο cold start. Τι είναι αυτό? Ανάβει στον κινητήρα και είναι τα, πρώτα πέντε λεπτά ε, ψυχρή κίνηση που είναι πάρα πολύ ψηλέ οι ε, εκπομπές. Και ε, αυτές μετρώνται, παρακολουθούνται και στην πραγματική οδήγηση αλλά δεν αξιολογούνται, δεν συνυπολογίζονται. Αλλά τα πρώτα 300 λοιπόν δευτερόλεπτα θα πρέπει να συνυπολογίζονται και η ψυχρή κίνηση στη συνολική μέτρηση των εκπομπών. Το βασικό ερώτημα που θα έπρεπε να απαντήσουμε στην ψυχρή κίνηση είναι πώς θα τα μετρήσουμε αυτά τα πέντε λεπτά και πώς, πώς θα τα συμπεριλάβουμε δηλαδή, γιατί αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης. Κοιτάξαμε διάφορες μεθόδους και τελικά καταλήξαμε στις πιο αξιόπιστες ή στην πιο αξιόπιστη. Και αυτό την ονομάζουμε κανονική πρόσθεση ε, των πέντε πρώτων λεπτών. Δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε ε, στη μέτρησή μας συν 300 δευτερόλεπτα. Ε, που θα πρέπει να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ όμως θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Σε αντίθεση με διάφορες φήμες που κυκλοφορούν και φτάσαν και στα δικά μας αυτιά, δεν είναι ένας τρόπος να διαλυθούν, να, να, να ενσωματωθούν ε, ε, αυτά στην οδήγηση στην πόλη. Όχι, τα μετράμε ξεχωριστά. Ξεχωριστά μετράμε ε, την οδήγηση στην πόλη που είναι και πιο ρηπαίνουσα και ξεχωριστά μετράμε το σύνολο της οδήγησης. Γιατί βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη ότι ρηπαίνουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα κατά την οδήγηση στην πόλη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που μελετήσαμε είναι η μέθοδος του ΕΚΟ, αν τα γνωρίζετε περισσότερα. Είναι ξεχωριστός υπολογισμός της ψυχρής εκκίνησης και της λειτουργίας του κινητήρα ε, ε, σε θερμό, ε, της λειτουργίας με θερμό κινητήρα Είναι περίπλοκοι αυτοί οι υπολογισμοί. Και είχαμε μια απόκληση της τάξης 7 με 46 χιλιόμετρων. Οπότε δεν υπάρχει ε, δυνατότητα ε, να μετρήσουμε την απόσταση ε, της ψυχρής εκείνης. Γι' αυτό μετράμε το χρόνο. Τα πέντε πρώτα λεπτά. Δηλαδή από, από, αρχίζοντας από μηδενική βάση, από τη στιγμή που ανάβει ο κινητήρας. Ε, επίσης μελετήσαμε και τη θερμή κίνηση. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που βγάλαμε από το σκάνδαλο των εκπομπών. Ε, λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα εκπέμπουν περισσότερα καύσα αέρια ε, με θερμό κινητήρα. Παρόλο που αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη λογική ούτε από τη φυσική, θα πρέπει και μία μελέτη, μία δοκιμή μάλλον να γίνεται με θερμό κινητήρα. Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι ε, αυτό που λέγεται regeneration event, δηλαδή ε, ανανέωση, καθαρισμού ας πούμε, αυτοκάθαρσης του, του αυτοκινήτου με διάφορα συστήματα, με φίλτρα, με ε, ε, Έχουμε λοιπόν ένα παράγοντα, ένα πολλαπλασιαστή δεν θα μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είναι ένας ακριβής τρόπος και αξιόπιστος να μετρηθούν και αυτά τα στοιχεία. Τέταρτον, τα ευρυδικά αυτοκίνητα. Ήταν επίσης σαφές ε, στο μυαλό μας και αυτό για το πώς συμπεριφέρονται τα υβριδικά αυτοκίνητα σε πραγματική οδήγηση. Είχαμε και διάφορα διλήμματα για το μέθοδο αξιολόγησης γιατί δεν είναι πάρα πολύ ακριβείς οι ε, σημερινές μέθοδοι. Επιλέξαμε μια άλλη μέθοδο ε, που μετράει και το διοξίδιο του άνθρακα και τα ε, οξύδια του αζότου. Και ένα τελευταίο που αξίζει να τονίσουμε είναι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, COC, Certificate of conformity. Προτείνουμε να γίνει υποχρεωτική η πληροφόρηση ήδη από τώρα για τους παράγοντες συμμόρφωσης για τον κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τριπλό στόχο. Πρώτον, αυτό, ο πρώτος στόχος είναι η διαφάνεια για να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, ε, να ξέρουν πόσο καλές ή κακές επιδόσεις έχει το κάθε όχημα. Ε, δεύτερον, αυτό μπορεί να δώσει και κίνητρα ε, στους κατασκευαστές για να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα αυτοκίνητα. Και τρίτον, ε, υπάρχει ένα στοιχείο σύγκρισης των αποτελεσμάτων που μας δίνουν οι κατασκευαστές με τα αποτελέσματα που παίρνουν από τις μετρήσεις ή ανεξάρτητοι οργανισμοί που τις διεξάγουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο για όλους και το τελευταίο για την προφόρηση για τον παράγοντα συμμόρφωση είναι ένα μέτρο που ενισχύει πολύ την ε, διαφάνεια. Και επειδή έχω περάσει το χρόνο μου κατά δυόμιση λεπτά, να σταματήσω εδώ και αν έχετε ερωτήσεις, αν ανέφερα κάτι επιγραμματικά και δεν το κάλυψα διεξοδικά, ρωτήστε με και θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Παρακαλώ. Κυρία Ανταλή, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις συνεκτικές πληροφορίες που μας έδωσε για το τι προτείνεται. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματικά τεστ στο δρόμο για να ελέγξουμε τις εκπομπές και επίση είναι πολύ θετικό να έχουμε μια διαδικασία που θα μπορεί να μετρά με ακρίβεια τις εκπομπές και να διασφαλίζει ότι τα πρότυπα της ρήπαν γίνονται σεβαστά στον πραγματικό κόσμο. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν το θέμα των σωματιδίων, στο οποίο αναφερθήκατε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό που η Κομισιόν προσπαθεί να εισαγάγει μέτρηση των σωματιδίων μέσω του φορετιού συστήματος μέτρησης εκπομπών, του ΠΕΜΣ, όμως ε, δεν έχω καταλάβει αν θα μετρήσουν ε, αυτά τα συστήματα όλα τα σωματίδια και τα κλάσματα. Ε, γιατί όπως έχουν τώρα τα πράγματα, εξακολουθεί να μπορεί να υπάρχει ένα κενό που μπορεί να γίνει αντικείμενο κατάχρησης από τους κατασκευαστές, ε, αν παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια σειρά μικρότερων σωματιδίων που δεν θα μετρηθούν. Έτσι λοιπόν, Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν αν ε, το σημερινό όριο ε, των σωματιδίων και ο εξοπλισμός ε, των ΠΕΜ μπορεί να μετρήσει τα σωματίδια όλων των μεγεθών ή κάποια θα μείνουν εκτός ρύθμισης. Και ποια είναι τα σχέδια της Κομισιόν έτσι ώστε και τα πιο επικίνδυνα και μικρότερα σωματίδια να μετρηθούν αποτελεσματικά. Και το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με τις συσκευές αναστολής. Στο εκτιμώντας 23 ε, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να απαντήσουμε σε αυτή την κατάχρηση των συσκευών. Όμως, καθώς οι εθνικές ε, ορχές ε, εξετάζουν εναλλακτικές μέτρησης, ή τελικά ε, τι σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αρχές θα εφαρμόζουν καταλήλως τους σημερινούς κανόνες. Επίσης, να ρωτήσω, η Κομισιόν θα εφαρμοζουν καταληλως του σημερινους κανονες εναρμονισμένους κανόνες για τις συσκευέ Ανατολής και αυτό θα είναι μέρος ε, των τεστ εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες και θα ελέγχεται και από τις αρχές έγκρισης ε, τύπου. Η Κομισιόν ουσιαστικά θα υιοθετήσει και τεχνολογία εχμής για αυτές τις συσκευέ. Ευχαριστώ κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εξηγήσεις αυτές. Έχω δύο τεχνικά ζητήματα και ένα διαδικαστικό. Καταρχήν, μια ερώτηση για τα σωματίδια και για τα φίλτρα. Αν με έχουν ενημερώσει σωστά, τα φίλτρα δεν ε, είναι ευαίσθητα προς τη θερμοκρασία. Δηλαδή λειτουργούν, ε, είτε είναι ψυχρός είτε θερμοστατινητήρας, απλώς λειτουργούν ως φίλτρα. Γιατί να κάνουμε μια διάκριση δηλαδή μεταξύ ψυχρού και θερμού κινητήρα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το συντελεστή συμμόρφωσης και ξέρουμε τι εννοούμε όπως και τον αποκαλούμε ότι επιτρέπουμε στα αυτοκίνητα να εκπέμπουν 50% περισσότερο από τα νόμιμα όρια, αν μιλάμε για 1,5. Με τα πέμ τα συστήματα μέτρησης εκπομπών και την μία ακριβή, αυτό σημαίνει ότι αν ε, χρησιμοποιήσεις το συντελεστή 1,5, Δηλαδή, σε αυτό σημαίνει ότι πιστεύετε ότι αυτά τα PEMS, τα φορητά συστήματα μέτρηση εκπομπών, ε, δεν εξυπηρετούν το στόχο, γιατί είναι ακριβή κατά 50%. Καλά το ερμηνεύω. Και αυτό είναι ένας λόγος που επιλέγεται το συντελεστή 1,5. Δηλαδή, ε, τελικά είναι ακριβή μόνο κατά 50% αυτά τα φορητά συστήματα μέτρηση εκπομπών σε ό,τι αφορά τα σωματίδια και σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις, ε, ομάδες, τις συναντήσεις ομάδας εργασίας ε, για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Πριν δύο εβδομάδες λάβουμε από την Κομισιόν τον κατάλογο των συμμετεχόντων, το όνομά τους και ποια οργάνωση εκπροσωπούν. 18 Μαΐου, 6 Ιουνίου και 8 Δεκεμβρίου φέτος ε, λαμβάνουν χωρές συνεδριάσεις και ο αριθμός των εκπροσώπων από τη βιομηχανία ήταν πάνω από 50% ε, σε όλες τις συναντήσεις. Ε, είχαμε ουσιαστικά 28-29 άτομα στα 45, στα 49 και διάβασα στον κατάλογο συμμετεχόντων ότι τα κράτη-μέλη έλειπαν σε μεγάλο βαθμό, ότι είχαμε μόνο εκπροσώπους από 2-3-4 κρατημέλη. Καθώς ε, αυτή η δουλειά είναι ιδιαίτερα πολιτική, περισσότερο από τεχνική. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί σε αυτές τις συναντήσεις της ομάδας εργασίας πάνω από το ίμιση των συμμετεχόντων είναι εκπρόσωποι του κλάδου. Σας ευχαριστώ, κύριε Σέικχαουτ. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση επίσης έχει να κάνει με το συντελεστή και με διόρθωσαν στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων, Επομένω, Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τη σωστή ορολογία. Εδώ δεν μιλάμε για συντελεστή συμμόρφωση του 1,5 για τα οξύδια του εζώτου, τώρα μιλάμε για σωματίδια. Όμω προσπαθώ να ακολουθήσω ότι παρακολουθήσατε, ότι χρειαζόταν ένα συντελεστή για να μετράμε τι ανακρίβειε του 0,5, τη τάξη του 0,5. Αλλά τελικά Καταλήγουμε στο ίδιο, το 50% των ορίων ε, ουσιαστικά ε, μπορεί να μην λευθούν, να ξεπεραστούν. Τώρα είτε το αποκαλείται αυτό συντελεστή ανακρίβειας, είτε συντελεστή συμμόρφωση, αλλάζεται το όριο που έχουμε συμφωνήσει στη διαδικασία συνομοθέτησης. Και με αυτό η βιομηχανία. μπορεί να εκπέμπει περισσότερο από αυτό που είχαμε συμφωνήσει εμείς ως συνομοθέτες. Ε, τελικά καταλήγουμε στο 2,50% παρόλο που δεν είναι τώρα αυτό συντελεστή συμμόρφωση και επομένω δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή τεχνικό λόγο γιατί προσθέτοντα ένα φίλτρο θα φτάσετε στα κατώτατα όρια. Τώρα λοιπόν μπαίνετε σε μια πολύ τεχνική συζήτηση με πάρα πολλού εκπροσώπου τη αυτοκινητοβιομηχανία σε σχέση με την ανακρίβεια των μετρήσεων PEMS, αλλά τελικά έχουμε μια απλή απόφαση. Θα εφαρμόσετε το φίλτρο, ναι ή όχι. Γιατί δεν το ξανακάνουμε όλο αυτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ποια κράτη-μέλη σα εξαναγκάζουν να πάτε προ αυτή την κατεύθυνση, θα ήθελα να μα το πείτε αυτό γιατί και πάλι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση η οποία ουσιαστικά λιώνει τα πρότυπα στα οποία συμφωνήσαμε ενώ δεν υπάρχει τεχνικός λόγος απλώς πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το φίλτρο είναι τόσο δύσκολο, δεν νομίζω να μας διαφωτίσετε παρακαλώ και θα θεωρήσω δεδομένο στη συνέχεια ότι δεν θα συζητήσουμε τη συντελεστή συμμόρφωση σε αυτή την περίπτωση του 50%. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Δεν το αναφέρεται καθόλου τη διαδικασία για τις κατευθύνες γραμμές για τις διατάξεις αναστολής. Πώς προοδεύουμε και πώς γίνεται αυτή η πρόοδος, αλλά και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πέφτουμε στην ίδια παγίδα. Δηλαδή ορίζουμε όλα τόσο πολύ σε τεχνικές επιτροπές και αν κάτι τελικά διαφέρει ελαχίστως δεν είναι πλέον συσκευή αναστολής. Γιατί ξέρουμε ότι τώρα υπάρχει μια συζήτηση μετά από 22 ε, λεπτά δεν είναι ε, συσκευή αναστολής ή αν έχουμε θερμοπαράθυρο. θα μας πείτε, θα μας πούν στη συνέχεια δεν έχει οριστεί, δεν είναι λοιπόν διάταξη αναστολής. Υπάρχει κάποιος τεχνικός ρόλος που θα ε, έχουμε ένα λογισμικό που θα λειτουργεί και κατόπιν θα σβήνει. Τέλο πάντων, αυτό που με ανησυχεί είναι να μην ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα, να έχουμε πλήρε λεπτομέρειες, πάρα πολύ τεχνικές και τελικά απλώ να βοηθήσουμε τον κλάδο στο να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Γιατί σε αυτές τι κατευθυρίες γραμμέ θα λένε Α, ό,τι δεν υπάρχει εκεί δεν είναι αυτό συσκευή αναστολής». Έτσι λοιπόν, να του βοηθήσουμε να μας ξεγελάσουν εκ νέου. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αυτό έχει σχέση με τη Συμφωνία για το Κλίμα και ε, το ρόλο που πρέπει να έχουν όλοι. Τώρα μιλάμε για ε, συστήματα μέτρησης που υπάρχουν, που κυκλοφορούν στην αγορά και το γνωρίζουμε. οι συσκευές PEMS πραγματικά δεν είναι επαρκείς για τη μέτρηση ε, σε πραγματικές ε, συνθήκες οδήγησης, ούτε για το οξύδιο του ε, αζότου, ούτε για το διοξίδιο του άνθρωπου. Και μιλάμε για ένα συντελεστή μισό, σε σχέση με το 1,5. Αναφέρθηκαν και άλλοι προηγουμένως σε αυτό η σημερινή γενιά ε, οργάνων PEMS μπορεί να ε, ανταποκριθεί γιατί έχει ακρίβεια μέτρησης μέχρι 0,3. Αυτά θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην τρίτη δέσμη. Στην ομοθεσία για τις ε, συνθήκες σε πραγματική οδήγηση Ε, έχουμε υποσχεθεί όλοι ε, ότι θα, θα πρέπει να θεσμευτούν όλοι οι κλάδοι να κάνουν αυτά που τους αναλογούν, συγκεκριμένη περίπτωση για τις ε, πραγματικές εκπομπές. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπένστον. Ευχαριστώ. Να δώσω συνέχεια σε αυτό που είπατε. Νομίζω ότι καλό να λέμε τα σίκα σίκα όταν μιλάμε για το παράγοντα συμμόρφωση 1,5. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που ήθελα να θέσω απευθεία είναι ότι ω προ τη διαδικασία. Γιατί και πάλι έχουμε εκτίμηση τη Επιτροπή για το βαθμό ανοχή σε σχέση με τι ισχύουσε τεχνολογικέ διαδικασίε. Πολύ ε, μακριά από το βαθμό συμμόρφωση που θα θέλαμε και στον οποίο θέλουμε να καταλήξουμε. Η εκτίμηση τη Επιτροπή είναι κάτι γύρω στο 30% με του εξοπλισμού PEMS. Το φορητό μηχανισμό υπολογισμού των εκπομπών. Πώς καταλήγεται σε αυτό το 1,5%. Και όπως ακούσαμε από την ε, βιομηχανία των καταλυτικών κινητήρων, υπάρχει η εκτίμηση για το ένα, για μονάδα. Ποια είναι η δική σας αιτιολόγηση. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Δεύτερη ερώτηση για τη διαδικασία της ψυχρής κίνησης. Γιατί χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα Γιατί χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα και ε, πρέπει να φτάσουμε στο μηδέν. Δεν είναι μεγάλη η χρονοθυρίδα που παρέχεται. Δεν είναι μεγάλος ο αντίκτυπος αυτής της ε, εκκίνησης. Ε, εδώ για τα μικρά σωματίδια. για τα σωματίδια αυτά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υγεία. Το θέμα είναι να δοθούν κινήτα στους κατασκευαστές για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα μίζωνα, ε, τα, για να αντιμετωπίσουν τα μείζωνα προβλήματα, δηλαδή τα σωματίδια που πραγματικά ε, μπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό και δημιουργούν ε, μακροχρόνια προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριο Τούρμες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θυμάμαι πολύ καλά όταν μας επισκέφθηκαν οι υπεύθυνοι της ε, εταιρεία για το gate. αυτό το, το σκάνδαλο που πραγματικότητα ένα σκάνδαλο diesel. Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το τι θα γίνει με τη διαδικασία των δοκιμών σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση. Και η EPA τότε μα είχε πει το ακριβώ αντίθετο από αυτό που λέτε εσεί. Σήμερα Εάν ορίσουμε τα πάντα καταλεπτός, ανοίγουμε την πόρτα στην εξαπάτηση, την ε, αλλίωση των κύκλων και τους μηχανισμούς αναστολής. Γι' αυτό η Αμερικανική EPA έχει εντελώ, ε, απόλυτη διακριτική ευχέρεια για το τι θα επιλέξει. Εδώ κάνουμε το Εδώ λοιπόν γι' αυτό κάνουμε τα ακριβώς ε, αντίθετα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι λεπτομέρειες ορίζονται για να μην, μπορεί, να μην μπορούν οι αυτοκινητοβιμηχανίες να ξαπατήσουν το σύστημα. Εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την Audi. Και πάλι έχουμε την πολύ ωραία ε, κατάσταση να έχουμε τις αρχές της Καλιφόρνιας να εντοπίζουν τις δικές μας ε, εξυπνάδες και δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες, χιλιάδες, ελπίζω όχι δις τέτοιων οχημάτων κυκλοφορούν στην Ευρώπη και η Επιτροπή τηρήσε γηχθείως. Δεν βλέπω καμία αντίδραση της Επιτροπής για την Audi. Ενώ οι αρχές της Καλιφόρνιας έχουν πει ήδη πολλά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εάν είσαστε σε επαφή με την Καλιφόρνια, τι σκοπεύετε να κάνετε και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω να ζητάει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή της Απαντήσεως. Όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν εκπλήσωμαι από τα σχόλια και από τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν. Ε, στη συζήτηση αυτή βλέπω σε μεγάλο βαθμό να δημιουργείται ένα κλίμα που έχει σχέση και με το συζήτηση που είχε γίνει για το RD2. Είχαμε συζητήσει διαφορετικά πράγματα. για τα τεστ σε πραγματικές συνθήκες. Εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε τις ε, καλύτερες γνώσεις που μπορούμε να έχουμε, το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό διαφάνειας και την τεχνική δουλειά της Επιτροπής μαζί με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καθώς και τους εκπροσώπους των βιομηχανιών, των ε, αυτοκινητοβιομηχανιών και των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει προτάσει που να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και τι δοκιμέ συνθήκη πραγματική οδήγηση. Γι' αυτό λοιπόν για τα σχόλιά σα και δεν ξέρω αν θα, καταφέρω να τα καλύψω όλα. Πρώτα απ' όλα τα σχόλια για τα σωματίδια. Εδώ είναι εύστοχη ερώτηση και συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να μιλάμε μόνο για 23 νανό ε, μόνο για 23 ε, νανομονάδες ε, σωματιδίων. Έτσι κι αλλιώς το θέμα άρχισε να συζητιέται πριν από δύο χρόνια στη Γενέβη, σε τεχνικό επίπεδο. Έχουμε ήδη προχωρήσει στο πώς ε, το εξετάζουμε και μην ξεχνάμε ότι οι βάσεις τα ήδη πριν από λίγο καιρό μόλις. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε και σε πόσο καιρό ακόμη, γιατί έχουν περάσει μόλι δύο χρόνια, αλλά συνεχίζουμε. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει το ε, να ορίσουμε πρώτα το πραγματικό μέγεθος των σωματιδίων, έστω και σε νανόμετρα. Ε, εδώ το άλλο θέμα είναι το τι κατευθυντήρια γραμμή θα δώσουμε. Ε, Δεν έχω ακόμη οριστικό αποτέλεσμα, αλλά επειδή την ερώτηση την έφεσαν πολλοί βουλευτές θα προσπαθήσω να απαντήσω. Έχουμε εργαστεί για τη γενική κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε όχι μόνο εμείς από τη δική μου ομάδα, αλλά το σχέδιο των συστάσεων το έχουμε δει και με τους συναδέλφους από την επιστημονική ομάδα Έχουμε δει ποια είναι η νομοθεσία που ισχύει στι ΗΠΑ και έχουμε δει το τι στοιχεία έχουμε από την πραγματικότητα. Δηλαδή περιπτώσει συγκεκριμένε ε, συσκευών αναστολή, τι οποίε έχουμε δει να διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Δεν σκοπεύουμε, όπω είπατε προηγουμένω, να αλλάξουμε του βασικού κανόνε για τι συσκευέ αναστολή. Θεωρούμε ότι η νομοθεσία όσο έχει τώρα είναι αρκετά σαφή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι όλη η διαδικασία από τις αρχές έγκρισης τύπου ολοκληρώνεται με τον τρόπο, με τον δέοντα τρόπο. Εδώ λοιπόν κοιτάζουμε να μην υπάρχουν παραθυράκια στο νόμο. Να μην γίνεται αξιόλογηση από τον ένα με τον ένα τρόπο και από τον άλλο με τον άλλο. Θέλουμε συγκεκριμένου κανόνε λοιπόν για τι διαδικασίε, διότι οι κανόνε, όπω είπα προηγουμένω, θεωρούμε ότι είναι αρκετά σαφεί ω προ τι απαγορεύσει, τις, ε, ε, τους αποκλεισμούς και τις εξαιρεσει. Έχουμε επίσης έναν κατάλογο με ενδεχόμενες ε, συσκευές αναστολής, ορισμούς, παραμέτρους, έναν ανοιχτό κατάλογο που βεβαίω δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί με τα αποκύματα τη μηχανική στο μέλλον. Εμεί δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε τώρα. Αλλά προχωρούμε σταδιακά για να έχουμε μια γενική κατεύθυνση έτοιμη στο τέλος της χρονιάς. Και οι στρατηγικές για την προστασία θα περιληφθούν όπως έγινε στη δεύτερη δέσμη και στην τρίτη και τέταρτη, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι συσκευέ αναστολή να, ως τέτοιες να ορίζονται και όλες εφόσον είμαι. Ως προς το πόσο ευαίσθητα είναι τα φίλτρα και τις θερμοκρασίες, Θα ζητήσω από τον ε, συνάδελφο που είναι ειδικό ε, στα θέματα αυτά να σας εξηγήσει πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται. Αλλά πρώτα απ' όλα για το περιθώριο του παράγοντα συμμόρφωσης. Αυτό που είπα και στην αρχή ισχύει. Αν δεν είχαμε συζητήσει για τα δεύτερη δέσμη, κανείς δεν θα ευνηδιαζόταν αν υπήρχε ένα περιθώριο, τέλος πάντων ε, μια, ένα περιθώριο ενοχής για το πώς μετράμε τις σε τι μονάδες και τον, ε, τα μεγέθη στα οποία μετράμε τις εκπομπές συνθήκης πραγματικής ε, οδήγησης. Τώρα θέλετε να το ονομάσετε παράγοντα συμμόρφωσης, το ονομάζουμε έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν συζητήσαμε αυτό διεξοδικό στις αρχές τη Ο εξοπλισμός είναι τέτοιο που μπορεί να έχει καλύτερα ή χειρότερα αποτελέσματα και δίνει διαφορετικά αποτελέσματα σε μία διαδρομή ή σε μια άλλη. Εξαρτάται πού τοποθετείτε. Αυτή είναι ακριβώ και η φύση του εργαλείου που χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, ρωτάτε κύριε Γερμπράντη εάν ο εξοπλισμό είναι κατάλληλος. Ναι, έχουμε κάνει μελέτες επί τριετία με το κοινοκέντρο για τα PEMS. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μετρώνται, όμως ο εξοπλισμός όσο έχει σήμερα δεν είναι και τέλειος. Το θέμα είναι ότι έχουμε λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε συμπεριλάβει, διότι με το 0,5 έχουμε κάνει σύγκριση των επιδόσεων από εργαστήριο σε εργαστήριο Ε, σε εργαστηριακέ συνθήκε έχουμε λάβει υπόψη την τάξη μεγέθου μέτρηση των ΠΕΜΣ, αλλά δεν έχουμε λάβει υπόψη τι πραγματικέ συνθήκε οδήγηση, ε, το πώ ε, καταναλώνεται τα καύσιμα, το ότι υπάρχουν διαφορέ από οχήματα σε οχήματα. Αυτό είναι ένα περιθώριο που θα πρέπει λοιπόν να το προβλέψουμε, αλλά δεν έχει να κάνει με τα ρυθμιστικά όρια. Είναι αυτά που είναι. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε 1,3 ή 1,2 φέτος του χρόνου. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τις συνθήκες, τους παράγοντες συμμόρφωσης. Ε, ελέγχουμε και άλλα στοιχεία, όχι μόνο τον εξοπλισμό αυτό καθεαυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια συγκεκριμένη εξήγηση και δεν είναι η Επιτροπή που είχε την ε, έμπνευση αυτή με τεχνικές δικές της γνώσεις. Επί τριετία μελετάτε το θέμα. Οι παραγωγοί αυτοκινητοβιομηχανίες μας λένε ότι υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να μετρήσει κάτω του 1,5. Αλλά ε, σίγουρα υπάρχουν τέτοια συστήματα μέτρησης, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανακρίβειας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στοιχεία που επιστημονικά να είναι εύρωστα και τα επιχείρηματά μας να υποστηρίζουν την τελική μας επιλογή. Δεν θέλαμε να πηγαίνουμε στη μέτρηση κάτω τη μονάδα, α πούμε, ή το, να δεχτούμε το ποσοστό πάνω το 300. Αυτά ε, επιλέξαμε γιατί ήταν τα, τα πλέον κατάλληλα κατά την άποψή μα. Αυτά ισχύουν σήμερα και γι' αυτό θα φροντίσουμε να νομοθετήσουμε για τη μέτρηση των πέμψη καταλήλω. Ω προ την ερώτηση για τη διαδικασία και πώ οργανωθήκαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ως συνήθως, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν ευρεία παρουσία. Υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να έρθουν αν θέλουν. Ναι, αν θέλουν οι πρόσωποι των κυβερνητικών οργανώσεων να προσέλθουν πολλοί άριθμοι, τόσο το καλύτερο. Δεν τους εμποδίζουμε. Η διαδικασία είναι τελείως ανοιχτή. Ο καθένα μπορεί να πάρει μέρος στις συναντήσει. Τους προσκαλούμε όλους αλλά δεν ξαναγκάζουμε και κανέναν να έρθει. Το θέμα είναι διαφορετικό. Ότι πρέπει να διαχειριστούμε τι συναντήσει με τρόπο κατάλογο, να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι παίρνουν το λόγο για να εκφράσουν τι θέσει του και να μπορέσουν να λάβουν και απαντήσει. Και πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει. Ω προ τα σχόλια για την συμμετοχή δύο ή τριών μόνο κρατών μελών, μην ξεχνάτε και ένα πράγμα. Τα κράτη-μέλη συζητούν και το έχουμε συζητήσει και εξωδικώ ήδη τέσσερι φορέ στην πρότασή μα με τα κράτη-μέλη την μόνιμη, και στο επίπεδο μόνιμη επιτροπή όπου υποβάλλουμε προτάσει και τι συζητούμε με τα κράτη-μέλη. Οπότε προφανώ τα κράτη-μέλη είναι μέλη, μέρη τη συζήτηση αυτή. Τώρα αν είναι δύο ή τρία είναι άλλο θέμα. Ε, όσοι παίρνουν μέρο στην ομάδα εργασία είναι αυτοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερω ή μα βοηθούν να συντάξουμε τι προτάσει, τα κείμενα. Είναι αναπόσπαστο μέρο τη διαδικασία. Αλλά να είστε βέβαιοι, τα κράτη-μέλη ε, τηρούνται ενήμερα από την ε, αρχή την ίδια τη διαδικασία μέχρι το τέλο τη ε, στη λειτουργία αυτή τη Επιτροπή. για τα 30 δευτερόλεπτα. Εάν είναι πολλά ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ορισμού. Εκεί θα κρυθεί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον ορισμό. Έτσι ορίστηκε η συσκευή αναστολή, έτσι είναι οι κανόνε. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για τι υπερβολικά πολλέ λεπτομέρειε ή το αντίθετο. Και το κατά πόσο είμαστε σε θέση να κάνουμε ανεξάρτητε δοκιμέ. Συμφωνούμε απολύτω μαζί σα. Το πρόβλημα είναι, όπω γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η νομοθεσία ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η Επιτροπή έχει περιορισμένε αρμοδιότητε. Δεν μπορεί να αλλάξει όλου του κανόνε, γι' αυτό προτείνουμε την νομοθεσία για την έγκριση τύπου. Εάν υπήρχαν διαφορετικέ δοκιμέ, δοκιμέ τελείω διαφορετικέ, δοκιμέ ευνηδιαστικέ ή δοκιμέ για την ε, ε, κατηγορία τύπου, αυτά είναι διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Αν αποφασιστεί να, κάνετε, να αλλάξουν οι κανόνε, αυτό θα το αποφασίσουν και θα κάνουν τα σχετική πρόταση και διαδικασία Συμβούλιο, ε, Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Για το τεχνικό τμήμα τη ερώτηση ο λόγο της συνάδελφου. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι ευνηδιάστηκα λίγο από τι ερωτήσει, διότι φαίνεται να υπάρχουν αρκετέ παρανοήσει για το τι μπορούν να κάνουν τα φίλτρα καθαρισμού των σωματιδίων και τι δεν μπορούν να κάνουν. Να εξηγήσω, όντω υπάρχει ένα φίλτρο που κατακρατά, όμω εάν ο κινητήρα ε, εκπέμπει πάρα πολλά, το φίλτρο θα κατακρατήσει κάποια, κάποια άλλα θα διαφύγουν. Επιπλέον, πραγματικά εκπλήσωμαι που έχετε πληροφορίες ότι τα οχήματα του GPF είναι κάτω του δεκαπλάσιου, του ενδεκαπλάσιου. Ε, διότι ακόμη υπάρχει, και αν υπάρχει μεγάλη φόρτωση ή οι δοκιμές γίνουν σε, στο 0, στη θερμοκρασία μηδέν του μηδενός θα τετραπλασιάσουμε κατευθείαν τον όγκο. Αν τα συνδυάζετε τώρα αυτά με δεδομένα που έχουμε για βαριά καύσιμα, καύσιμα που μπορεί να κυκλοφορούν περιορισμένα στην αγορά, όχι στη βασική δηλαδή αγορά, στο 5% των βαρέων της ε, ευρωπαϊκής αγοράς, αλλάζει πάλι ο συσχετισμός. Δηλαδή ένα όχημα που υποτίθεται ότι είναι πολύ κάτω του ορίου, μπορεί στην πραγματικότητα να το έχει υπερβεί. Να έχει υπερβεί τον ε, εαυτό του και το όριο του γύρω 6. Αυτός είναι ο λόγος που είπαμε ας τα αφήσουμε αυτό. Θα κοιτάξουμε μόνο πόσο παραπάνω μετρά ο εξοπλισμός όταν μετράει ίδια πράγματα. Δηλαδή παίρνουμε το όχημα σε ένα εργαστήριο, πολλά όχηματα μάλλον στο εργαστήριο, πολλά σε διαφορετικά εργαστήρια και, και κάνουμε πολλές διαφορετικές μετρήσεις. Με 50% Βεβαιότητα. Το 30% που αναφέρατε εσεί ήταν για ένα εργαλείο που δεν ήταν κατάλληλο στην πραγματικότητα. Το εργαλείο αυτό σε χαμηλέ θερμοκρασίε έπαθε να λειτουργεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάζουμε την νομοθεσία μα σε κάτι που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλε τι περιπτώσει, σε όλη τη διαδικασία των ε, συνθήκων μέτρηση πραγματική οδήγηση. Αυτά προ στιγμή. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις δεν απαντήσατε για την Άουμπι. Αυτό που είπαμε τις αρχές της Καλιφόρνιας. Για το θέμα αυτό δεν είμαστε σε συνεννόηση με τις Αμερικανικές αρχές. δεν έχουμε συνεννοηθεί με το σχετικό συμβούλιο της Καλιφόρνιας. Όμως την EPA ε, θα ενημερωθούμε απευθείας εάν ε, προκύψει αυτό και θα σας πούμε τι έγινε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης. Ένσταση βάσει του άρθρου 106 για το ρόλο της ε, ενεργό ουσίας ε, βενταζόνης. Θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους και όλους τους, τους συνεργάτες να μας αφήσουν την ευκαιρία να συνεχίσουμε. Δεν έχει λήξει η συνεδρίαση. Παρακαλώ, εάν θέλετε να εξέλθετε, ησύχως, για να συνεχίσουμε. Ο λόγος στον εισηγητή, τον κύριο Πότς. Yes, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την γενοδορία τους ε, που αποχωρούν ησύχως από την αίθουσα. Να πω ότι έχω κουραστεί να φέρνω αντιρρήσεις, όμως ε, λυπάμαι. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά στην περίπτωση αυτή. Και πάλι εδώ συζητούμε την ε, αντίρρηση που έχει να κάνει με τον άρθρο 106 και την ανανέωση μιας δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται σε προϊόντα φυτοπροστασίας. Αυτή τη στιγμή συζητούμε το Μπέντεζον, το οποίο χρησιμοποιείται στη Γεωργία, έχει υψηλό, υψηλή δυνατότητα να φτάσει στα υπόγεια ύδατα και ουσιαστικά το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το Ενωμένο Βασίλειο και σύμφωνα και με δεδομένα από τον ίδιο τον ΕΤΟΥΤΑ, αυτή η κατάσταση συναντάται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης οι χημικές του ενώσεις είναι και ενδοκρινικές διαταράκτες. Η Κομισιόν και πάλι δεν σεβάστηκε ε, τον, ε, κανόνες, τον κανονισμό 1107-2007 σε σχέση με τα παρασιτοκτόνα. Ε, ουσιαστικά δεν σέβεται την αρχή της πρόληψης που έχουμε στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Κομισιόν ε, προτείνει ε, ουσιαστικά ε, να ανανεωθεί η έγκριση του πενταζών μέχρι το 2032 για 15 χρόνια παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει δεδομένα που να μας διαβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλές το μπενταζόν και ταυτόχρονα ζητά αυτά τα δεδομένα από τον ετούντα ο οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ασφάλεια αυτής της ουσίας. Αυτή η πρακτική ε, έχει ε, γίνει ε, έχει επικριθεί αρκετά, δηλαδή να δίνεται η άδεια κυκλοφορία στην αγορά στο προϊόν πριν να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Η απόφαση του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή σε σχέση με τις πρακτικές της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την έγκριση και τη θέση σε εμπορία των παρασυντοκτώνων καλεί την Κομισιόν να πάψει να χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία. Η Κομισιόν έχει δεχτεί την πρόταση του διαμεσολαβητή για πάρα πολλά θέματα που αφορούν αυτή τη διαδικασία, όμως ε, δεν, ε, και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι έχει αποτύχει να ακολουθήσει τη σύσταση του διαμεσολαβητή. Εδώ Για να σεβαστούμε την υφιστάμενη νομοθεσία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια θέση οι εγκεκριμένε ουσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι ασφαλείς ή να μην σέβονται τη σχετική νομοθεσία. Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εγκρίνονται δραστική, μια διαστική ουσία για 15 χρόνια πριν να έχουμε την αξιολόγηση των καταναλωτών και πριν να έχουμε μια αξιολόγηση έκθεσης ε, των ε, ανθρώπων στην ουσία αυτή, πριν να έχουμε διαβούλευση εμπειρογνωμόνων της ΕΦΣΑ σε ό,τι αφορά τα κατάλοιπα, την τοξικολογία, την οικοτοξικολογία κτλ. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι μπορούν να κατανοήσουν την αντίρρησή μου και την αποστηρίξουν και να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού η Κομισιόν και να παρουσιάσει μια νέα πρόταση όπου θα έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στους ομιλητές. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που τονίσαμε ότι πρόκειται για εκτελεστική πράξη, δηλαδή εμείς ως Κοινοβούλιο συμμετέχουμε έμεσα και όχι άμεσα και την πραγματική δουλειά πρέπει να την κάνει η Κομισιόν με το Συμβούλιο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, επειδή ασχολούμαι και με τη γεωργία και θέλω να το σκεφτούμε, το βασικό πρόβλημα είναι οι διτές αποφάσεις, τι εννοώ, όχι διτές ακριβώ αυτό το άσπρο μαύρο, το, οι διπολικέ. δεν, δεν μπορείς να πει ότι αυτό το χωριό είναι καλό ή το άλλο είναι κακό. Και μιλήσαμε για του ενδεχόμενου ενδοκρινικούς διαταράκτε που να δείτε ο καφέ πόσα τέτοια περιέχει. Τι θα κάνουμε, θα απαγορεύσουμε να πίνουμε καφέ. Δηλαδή, δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι μόνο το θέμα η δραστική ουσία, αλλά και πώ χρησιμοποιείται και η συγκέντρωση για το αν είναι κάτι φάρμακο ή φαρμάκι. Βεβαίω δεν μπορούμε να διαπλεκτιζόμαστε συνεχώς. Το πενταζόν χρησιμοποιείται στη Γεωργία μεν, ε, αλλά αυτό δεν ε, δικαιολογεί καθόλου την αντίρρηση. Μπορούμε δηλαδή να διαφωνούμε για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ή όχι, αλλά δεν δικαιολογεί την αντίρρηση. Υπάρχουν ε, και επιστημονικές μελέτες που μπορούν να πούν ότι η δραστική ουσία βεβαίως από μόνη της είναι ζυζανιοκτόνο και αυτή είναι η ιδιότητα των φυτοφαρμάκων ότι προστατεύουν κάποια φυτά και κάποια άλλα τα σκοτώνουν. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε κιόλα. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητήσουμε τη χρήση, αλλά αν είναι η χρήση συνετή, ορθή, σεβόμενη όλους τους περιορισμούς και τις διατάξεις, κατά την άποψή μας η αντίρρηση αυτή δεν ευσταθεί και δεν δικαιολογείται. Αυτά προς το παρόν και σύντομα. Δηλαδή απορρίπτω την αντίρρηση αυτή. Thank you very much. Ms. Gerling. Thank you, Chairman. I'm glad... Ευχαριστώ. Λέω κύριε Γκέρλινγκ. Χαίρομαι που ακούω τον ε, κύριο Πότσο να λέει ότι κουράστηκε ε, για αυτές τις ε, αντιρρήσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχω πει πολλάκις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες η Κομισιόν επειδή δεν μας αρέσει το περιεχόμενο των μέτρων. Ο κανονισμός PPP ε, προβλέπει να ασκεί η Κομισιόν τις αρμοδιότητές της ε, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν από διαδικαστική σκοπιά δεν θα πρέπει να φέρνουμε εδώ αντίρρηση. Νομίζω ότι συνεχίζοντας να κάνουμε κάτι τέτοιο, όπως κάπτουμε το έργο της Επιτροπής μας και κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι άνθρωποι να μας ακούνε και ξέρω αρκετούς που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, για το περιεχόμενο. Εγώ έχω ένα θέμα με μερικά στοιχεία του ψηφίσματος. Δεν θα αναφερθώ τώρα λεπτομερώς, απλώς θα αναφερθώ στα σημαντικά. Και κατά την άποψή μου νομίζω ότι δεν παραθέσατε σωστά το διαμεσολαβητή λέει ότι απευθύνθηκε στην Κομισιόν και είπε να χρησιμοποιηθεί αυτή τη διαδικασία της λογής δεδομένων και θα έπρεπε να λέει χρησιμοποιήστε τη διαδικασία περιοριστικά μόνο σε περιπτώσεις όπου αιτιολογείται λέει δεν σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτή τη διαδικασία, αλλά προσέξτε πώς τη χρησιμοποιείτε. Έτσι λοιπόν, είναι τέλος ανακριβέ να λέτε ότι είπε διαμεσολαβητής Σταματήστε. Επίση, λέει, δώστε προτεραιότητα στο να ζητήσετε οποιασδήποτε λυπής πληροφορίες πριν να λάβετε απόφαση για την έγκριση. Έτσι λοιπόν, πηγαίνω στο άλλο μου σημείο. Το ε, ε, συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Κομισιόν χρησιμοποιώντα αυτή τη διαδικασία έχει παραβιάσει τι διατάξει του κανονισμού PPP. Αυτό δεν ισχύει γιατί στην περίπτωση των πενταζών ε, τα μόνα δεδομένα που ζητηθήκαν να αφορούν τα τεστ που έχουν να κάνουν με ε, τρόπο δράσης ουσιών που αφορούν τις ενδοκρίνες και βάσει ουσιών που δοκιμάστηκαν σε αρουραίους εδώ. Θα έπρεπε να δούμε τα ενδιάμεσα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς ε, διαταράκτες, όμως τώρα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, συνεχίζεται αυτό το έργο, κανείς δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να γίνει, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε είναι οποιαδήποτε αίτηση να την παγώνουμε ε, περιμένοντας να τελειώσουμε τη δουλειά μας για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ουσιαστικά, αν αφήσουμε κάτι να περάσει, υποστηρίζουν κάποιοι, εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Ακόμη και αν ολοκληρωθεί η δουλειά για του ενδοκρινικούς διαταράκτε, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το προϊόν, υπάρχουν διαδικασίες που σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φοβόμαστε μια πραγματική έγκριση σε αυτό το σημείο, καθώς δεν έχουμε δεδομένα να πούμε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί νέα έγκριση. Δεν ισχύει σε αυτή την ε, περίπτωση. Μέχρι να έχουμε τα δεδομένα που αφορούν του ενδοκρινικού διαταράκτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ούτε μπορούμε να αποσύρουμε προϊόντα από την αγορά που είναι χρήσιμα και σε αυτό το στάδιο δεν ξέρουμε να δημιουργούν προβλήματα και απλώς θα υπερφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάλμπερν, ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ε, έχω έτοιμη την κρίση μου τώρα όπως πολλοί συνάδελφοι. Θέλω να ακούσω πρώτα την Κομισιόν να μας πει γιατί πήρε αυτή την απόφαση που πήρε. Thank you very much. Ευχαριστώ. Άουκεν. Σας ευχαριστώ που διαμαρτυρηθήκατε, κύριε Πότσο. Εμείς οι πράσινοι είμαστε μαζί σας. Και δεν έχουμε μόνο τα δεδομένα για τους μικρονικούς διαταράκτες. τους χάρη, για το θέμα της τοξικότητας, ούτε εκεί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και έχουμε μια αρχή της πρόληψης που είναι βασική στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Μεσολαβήτη δεν θα πρέπει να αφιζητηθούν εδώ. Λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πρακτική όταν εξακολουθούμε να ζητούμε δεδομένα. Και δεν ξέρουν όλες οι χώρες ε, ποια είναι η δουλειά του Ευρωπαϊκού Μεσολαβητή. Όμως ε, εδώ δίνεται αυτή η έγκριση για 15 χρόνια. Όταν εξακολουθούμε να μην ξέρουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της ουσίας. Νομίζω ότι εδώ υποσκάπτεται όχι μόνο υγεία των ανθρώπων αλλά ε, και της φύσης αλλά και εμπιστοσύνη στην Κομισιόν γιατί η Κομισιόν ξανά και ξανά εμφανίζεται αδύναμη σε ό,τι αφορά το σεβασμό των προτύπων, των νόμων, των ερχών. Και αυτό το βλέπουν και οι πολίτες μας και δεν μας εμπιστεύονται. Γιατί φαίνεται ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά τη δική μας νομοθεσία και τη δική μας αρχές. Ελπίζω λοιπόν να μπορούμε να έχουμε μια πλειοψηφία, γιατί βλέπω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Ο κύριος Σούλφ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ για ένα τέτοιο θέμα, ε, οπότε δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερο. Ε, μπενταζόν. Διαδικασία ανανέωση. Ημερομηνία ε, λήξη τη έγκριση 2007 Ιούνιο. Πρώτη συζήτηση για το σχέδιο. Το σχέδιο στο οποίο αναφερθήκατε με τα κράτη-μέλη και την Εθνική Επιτροπή έχει προηγηθεί και να θυμίσω πριν πω στις λεπτομέρειες ε, στις ότι η διαδικασία για την οποία ε, συζητούμε σε ενωσιακό επίπεδο για την έγκριση των ουσιών αυτών έχει να κάνει με το σημαντικό ρόλο των κρατών μελών στην εξουσιοδότηση των φυτογενομικών ε, ουσιών. εκφράστηκε μια σειρά από ανησυχίες για τους υδροφόρους ορίζοντες, τους ενδοκρινικούς διταράκτες, αλλά και άλλα οριζοντιότερα θέματα, όπως την ε, συμμόρφωση Για τα στοιχεία επιβεβαίωσης. Εδώ λοιπόν ε, παρακολουθούμε αυτά που λέει και η κυρία και ότι θα πρέπει για την εξοδότηση των ουσιών η Επιτροπή να σταματήσει να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους επιβιωτικά δεδομένα. Ο Ombudsman ε, στο πορίσμα του αναφέρθηκε στη χρήση των ε, στοιχείων αυτών επαλήθευσης βάσει των όσων έχουν ε, ήδη ισχύσει για την θέση σε εμπορία της οδηγίας 414. Ο Ombudsman κατέληξε ότι στην οδηγία 14, 41-14 91-4-14 δεν λέγεται ότι τέτοια είδους, τέτοια είδους δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν υπάρχουν νέες απαιτήσει κατά τη διαδικασία έγκρισης, ε, αξιολόγηση, μάλλον, δηλαδή μετά την υποβολή αίτηση από τον ε, Τουντά, ο οποίο δεν πρόλαβε την προθεσμία για να συμπληρώσει τα στοιχεία, ή όταν ένας υποψήφιο υποβάλλει τέτοια στοιχεία για δεύτερη ε, νέα, εφόσον προέκυψαν νέε επιστημονικέ γνώσεις κατά τη διάρκεια τη διαδικασία αξιολόγηση λαμβάνουμε προφανώ πολύ σοβαρά υπόψη την απόφαση, το πόρισμα του διαμεσολαβητή. Τώρα, δεύτερο σημείο. Ενδοκρινικοί διαταράκτε. Το λέω, αλλά δεν είναι σωστό. Η ΕΦΣΑ λέει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να ε, επιβεβαιώσουμε ότι το έξιν είναι η δράση του στοιχείου αυτού ε, ε, προκαλεί ενδοκρινικές διαταραχές. Τα Στοιχεία λοιπόν επιβεβαίωσης και ενδοκρινικές διαταραχές που προκαλεί, θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχει και δράση ε, που να προκαλεί ενδοκρινικές διαταραχές και πρέπει να αναχαιτιστεί, όπως λέει και η ΕΦΣΑ. Η αίτηση για τα επιπλέον στοιχεία ήδη έχει αποσταλεί στην ΕΦΣΑ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, προκειμένου να μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί, να κατηγοριοποιηθεί ως τοξική κατηγορία 2 το βενταζόν. Το, η ουσία μπενταζόνη έχει λοιπόν ταξινομηθεί βάσει των σχετικών ε, ε, κανόνων, όμως αυτή η κατηγοριοποίηση δεν έχει καθόλου προβλέψεις για την ε, αμοιβαία τοξικότητα. Εδώ λοιπόν Εδώ δεν προβλέπεται ειδική κατηγοριοποίηση για την ε, Βενταζόνη και ο ετών ή δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει Εδώ δεν ξέρουμε ε, κατά πόσον μπορεί να πιστοποιηθεί η δεν γνωριζε η δεν μπορουσε να γνωριζει εδω δεν ξερουμε κατα ποσον μπορει να πιστοποιηθει η σχέση της μεταζώνης με τις ενδοκρινικές διαταραχές. Έτσι κι αλλιώς στο σχέδιό μας φροντίζουμε να ζητήσουμε από τον ε, Τούντα να υποβάλει περιττέρω στοιχεία μέχρι το 2018 προκειμένου να τα αξιολογήσουμε. Ένα άλλο σημείο που εφήγει και έθεσε να αμφιβόλο το κατά πόσο είναι ασφαλή η ουσία έχει να κάνει με του υδροφόρου ορίζοντε. Κατά πόσο η βενταζόνη μπορεί να φτάσει στα υπόγεια ύδατα. Κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε και το οποίο υπόθηκε επανειλημμένος για το αν υπάρχει αντίκτυπος. Ο Ετών υπέβαλε αίτηση για τις διάφορες συνηθισμένες χαρακτηριστικές χρήσεις και η αξιολόγηση η αποτίμηση, η ενδυνάμει ρήπανση των υπογείων υδάτων βασίστηκε σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο μελέτης, το λεγόμενο focus model, το οποίο λαμβάνει υπόψη διάφορες, ε, διάφορες ε, συνθήκες των υδροφόρων οριζόντων και κλιματικές συνθήκες για να δούμε πώς επιδρά η βενταζόνη. Είναι πολύ λεπτομερές και διξοδικό το μοντέλο αυτό. Όταν οι υπεύθυνοι για τη μελέτη αντικτύπου, λοιπόν, για την αξιολόγηση κινδύνου έστειλαν τα στοιχεία στα κράτη-μέλη, φάνηκε ότι στα 7 από τη 9 ε, στοιχεία με 160 γραμμάρια ένα εκτάριο έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Όλες οι άλλες χρήσεις 160 γραμμάρια πάλι δεν προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες. για την έγκριση της ουσίας ήταν αρκετό μία ασφαλής χρήση να εντοπιστεί. Εμείς έχουμε φτάσει στις 9, έτσι κι αλλιώς. Έπειτα για την έγκριση της ουσίας απαιτείται από τα κρατη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ε, υπόγειων ε, υδάτων αλλά και των φυτών που περιέχουν, ε, στα οποία χρησιμοποιείται η πενταζόνη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να απορρίψουν την έγκριση από άλλο κράτος μέλος, ε, εφόσον υπάρχει μία αποδεκτός κίνδυνος για το περιβάλλον σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένα να ε, εφαρμόσουν την αμοιβαία αναγνώριση. Επειδή το σχέδιο είναι εμπιστευτικό, δεν ακολουθούσαμε τη δημοσιοποίηση των δεδομένων όπως έβλεπε ο κανονισμός 1107 του 1999 και επιπλέον βάσει του πορίσματος του, του Ombudsman δεν θέλαμε να αντικρούσουμε και στην αρχή της προφύλαξης. Γι' αυτό επιτρέψαμε την ανανέωση τη δραστική ουσία βενταζόνη, γιατί εντοπίσαμε ακριβώ όπω σα είπα τι ασφαλεί χρήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εφόσον μας απαντήσατε να δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγα δευτερόλεπτα θα μιλήσω εγώ μόνο. Θέλω να πω στους αξιότιμους συναδέλφους ε, και στον συνάδελφο από τον ΕΛΚ ε, ε, Εγώ δεν αντιλέγω ότι είναι χρήσιμη η ουσία αυτή για τη γεωργία. Καταλαβαίνω ότι κάποια μέρα μπορεί να εγκριθεί και να χρησιμοποιείται στη Γεωργία, αλλά δεδομένη τη χρήση τα τελευταία 15 χρόνια με τον τρόπο που γίνεται, χωρί τα στοιχεία και τα δεδομένα, δεν γίνεται. Για να ξέρουμε αν αυτή η δραστική ουσία είναι ε, ε, καλή ή όχι. Η, οχι ε, ασφαλης Και για την τζουλι Γκέρλινγκ τα παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη, μην νομίζεις. Εσύ λες ότι προ, ε, προτιμάς την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, το ρίσκο και εγώ την προφύλαξη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ε, καταλαβαίνω. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να την ευχαριστήσω που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μου. Και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θυμίζω ότι στις 8 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα, αύριο δηλαδή. Λήξη της απόψινής συνεδρίασης θα λέμε αύριο το πρωί στο καλό να πάτε.